Να ξεκινήσουμε λοιπόν την ακρόαση που έχει θέμα απόδοση και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εφαρμογής και ελέγχου του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και προτάσεις αναθεώρησης. Και να πω στους δύο παριστάμενους ε, βουλευτές ποιε είναι οι αποφάσεις που πήραμε χθε στην συνεδρίαση των συντονιστών. Θα είμαι πολύ σύντομο έτσι ώστε να ξεκινήσουμε με την ακρόαση. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με τις ειδικέ εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου ε, ορίστηκαν οι ομάδες που θα είναι οι συγκητές, το ΕΛΚ θα ασχοληθεί με τις τρεις ειδικέ εκθέσεις της, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Επίσης, σε σχέση με την ε, διοργανική συμφωνία για θέματα προϋπολογισμού και σε σχέση με τις ε, πέντε ε, μελέτες οι οποίες εκπονήθηκαν και παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση ορίστηκαν οι αρμόδιοι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής μας που θα παρακολουθήσουν τα θέματα. Εκτός από το σημείο 4 ε, που ε, επιφυλάχθηκε η σοσιαλιστική ομάδα να αναφέρει το όνομα του εισηγητού. Όσον αφορά την επόμενη μεταρρύθμιση της Eurojust και λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο μεταρρύθμισης το οποίο θα πρέπει να ε, υποβάλει ο Ορμόδιος Επίτροπος για την Όλαφ καθώς επίσης και την ακόλουθη συζήτηση στο Κοινοβούλιο λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη ότι η συζήτηση με την Όλαφ βάσει της οποίας έχει προβλεφθεί ακρόαση ε, για την 12η Ιουλίου με τον Επίτροπο Σεμέτα, λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν την απαραίτητη προτεραιότητα που αποτελεί για μας και μέσα στα πλαίσια ε, υγιούς και καλής συνεργασίας θα ε, συνεργαστούμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ βάσει του άρθρου 151 ε, και θα ε, γίνουν από κοινού λοιπόν οι συζητήσεις για την Eurojust έτσι ώστε να δούμε ε, κατά πόσον είναι δόκιμο να υπάρξει μια κοινή συνεδρία των Επιτροπών Ελέγχου του Προϋπολογισμού και ΛΥΜΠΕ. Επιβεβαιώθηκε η αποστολή του Ιουνίου στην Κροατία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και η Πατριτσόλα Μαρκοβέρο Κονσολίνο και Βάουγκαν θα είναι παρόντες στην Επιτροπή αυτή. Για την 1η Ιουνίου 2010 προβλέπεται ακρόαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και Επιτροπής των Προϋπολογισμών σχετικά με την αναθεώρηση του ε, δημοσιονομικού κανονισμού. Επίσης, οι ε, συντονιστές επέτρεψαν στον πρόεδρο και μόνο στον πρόεδρο, ε, ε, προς τον πρόεδρο της, των προϋπολογισμών ένα σχέδιο επιστολής προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Επίσης, 13 Ιουλίου έχουμε τον, την ακρόαση όπου ο εισηγητής κύριος Λιμπεράσκη θα ασχοληθεί με το θέμα της διαφάνειας των διαρθρωτικών ταμείων και των των διευθυντικών ταμείων. Επίσης, ε, αναφορά του κυρίου Αλάκη, ο οποίος ασχολήθηκε με, συμμετέσχε, μάλλον στην πρόσφατη επίσκεψη του Κοινοβουλίου στο Αφγανιστάν, στις εργασίες που έγιναν επιτόπου από την ε, Επιτροπή αυτή, στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Αρλέκη, θα γίνει συζήτηση για τους δωρητές, για τα χρήματα τα οποία έχουν ε, πάει προς το Αφγανιστάν είτε από διεθνείς οργανισμούς ε, είτε ε, από κράτη και που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ όσοι συμμετέσχουν σε αυτήν τη συνάντηση, σε αυτήν την αποστολή στο Αφγανιστάν διεπίστωσαν και ήταν παρόντες και δημοσιογράφοι ότι το 80 περίπου των χρημάτων που δόθηκαν δεν έφτασαν ποτέ ε, επιτόπου και δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Επίσης, επί του θέματος θα πρέπει οι σοσιαλιστές να ε, ορίσουν κάποιον ε, κάποιον εισηγητή ή κάποιον υπεύθυνο. Στα υπόλοιπα σημεία δεν έχουμε καμία απόφαση. Αναφέρθηκα λοιπόν σε όλες τις αποφάσεις που πήραν οι συντονιστές χθες. Παρακαλώ κύριε Άουντι, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας ευχαριστήσω που βάλατε στην ημερήσια διάταξη και το θέμα της αποστολής στην Κροατία. Όσον αφορά τώρα τις μελέτες, τον προγραμματισμό των μελετών αυτών, έχει ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο μελέτης ε, του, της περιμέτρου ελέγχου ε, του Κοινοβουλίου υπό το φως των αλλαγών της συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι καλό να έχουμε μια τέτοια μελέτη ε, στα πλαίσια της προσεχούς τριετούς αναμόρφωσης και νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουμε ακριβώς ποιες είναι οι νομικές εξουσίες που έχουμε όλοι μας, η μεν και η δε. Ωραία, μπορούμε να προχωρήσουμε στην, με την συζήτησή μας. Και έχουμε λοιπόν το σχέδιο εμείς διάταξης για την ακρόαση με θέμα απόδοση και αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου και εφαρμογής του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και προτάσεις αναθεώρησης. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παρισταμένους. Θα ακούσουμε ε, όλους με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή γιατί το θέμα της έρευνας είναι απόλυτα σημαντικό. Εδώ και πολλά χρόνια η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, όπως και το υπόλοιπο Κοινοβούλιο, αλλά κυρίως η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, ε, έχει ασχοληθεί ενδελεχώς με θέματα διαφάνειας του δημοσίου χρήματος. Το, τα, δημόσια ταμεία δίνουν μια εξαιρετική ευκαιρία ανάπτυξης πολιτισμού, έρευνας, ενίσχυσης του Πανεπιστημίου, κυρίως δε στα πλαίσια της ε, τρίτης ε, χιλιετίας να, να, να βοηθήσουν έτσι ώστε να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη συμβατή με το περιβάλλον. Ε, είναι γεγονός και το γνωρίζουμε ότι ένα τμήμα του δημοσίου χρήματος, των δημοσίων ταμείων δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Απ' την άλλη πλευρά γνωρίζουμε επίσης ότι οι πόροι των ε, ταμείων μας πολλές φορές χρησιμοποιούνται άσχημα ε, και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα πρόβλημα γιατί υποσκάπτει το μέλλον της Ευρώπης, το μέλλον της ανθρωπότητας, το μέλλον της πρόοδου. Η χρήση λοιπόν των ε, χρημάτων των Ευρωπαϊκών Ταμείων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπε και η Επιτροπή αλλά και ε, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα όσον αφορά τα ε, δημόσια, τα ταμεία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γεγονός ότι μέσα σε ένα περίπλοκο νομοθετικό πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο περίπλοκων και πολλαπλών κανόνων, η διαφάνεια είναι λίγο πιο δύσκολο να αποδειχθεί και αποτελεί συχνά πρόφαση αυτή η πολυπλοκότητα των ε, κανόνων για την ελλειπή ή εσφαλμένη χρήση των πόρων αυτών. Εμείς πλέον λέμε ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα των Ευρωπαϊκών Ταμείων για προσωπικό πλουτισμό. Αυτό άλλωστε ε, διακήρυξε και ο κύριος Λιμπεράσκη ε, όσον αφορά στην απαλλαγή του προϋπολογισμού 2007. Αυτό λέμε σαν Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ε, και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε όλοι οι πόροι να χρησιμοποιηθούν σωστά για προγράμματα έρευνας έτσι ώστε οι τελικοί αποδέκτες, δηλαδή οι πολίτες της Ευρώπης, να είναι ε, αυτοί οι οποίοι τελικά θα ωφεληθούν από τους πόρους αυτούς. Θα δώσω το λόγο ε, αμέσως στον πρώτο εισηγητή, Γενικό Γραμματέα της Ερευνητικής Κοινότητας ΕΑΡΤΟ, κύριο Κρίστοφερ Χάλ, τον οποίον ευχαριστώ ζητώντας του να μην ξεπεράσει τα 15 λεπτά που έχουν οριστεί για κάθε ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να έρθω εδώ σήμερα και να σας μιλήσω για θέματα με την εφαρμογή και την εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου. Υπάρχουν μερικά πράγματα εδώ που θα έπρεπε επιγόντως να προσέξουμε και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να παίξει σημαντικό ρόλο προκειμένου να βρει λύσεις και να βελτιώσει την κατάσταση. Πριν έρθω όμως αυτά, επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σας πω δύο λόγια για την, ε, τις οργανώσεις που εκπροσωπώ εγώ και την Ερατό γενικότερα. Πρόκειται για οργανώσεις που ασχολούνται με την τεχνολογία. Εκπροσωπούμε 350 τέτοιες οργανώσεις από ολόκληρη την Ευρώπη. Για να δώσω έναν απλό ορισμό, είναι οργανώσεις που ασχολούνται με την έρευνα και αναλαμβάνουν κυρίως εφαρμοσμένη έρευνα. Οι περισσότερες χρηματοδοτούνται από κυβερνήσεις, συνεργάζονται με κυβερνήσεις για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, πράγματα που σήμερα αποτελούν μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Ε, συγχρόνως ασχολούνται και με την ε, ανταγωνιστικότητα όταν συνεργάζονται με επιχειρήσεις τόσο μεγάλες όσο και μικρές. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε μερικές ε, από αυτές, αλλά υπάρχουν στη διαφάνεια έτσι κι αλλιώς και κάτω βλέπετε και κάποια νούμερα, τα οποία πιστεύω ότι σας δείχνουν ότι αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα του προγράμματος αυτού πλαισίου. 30% του προγράμματος αυτού ήταν για οργανώσεις ερευνητικές των πανεπιστημίων. Ας έρθουμε λοιπόν ε, λιγάκι τώρα στο σημερινό μας ζήτημα. Υπάρχουν διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την εκτέλεση, την εφαρμογή του 7ου προγράμματος πλαισίου. Πάντως, και άλλα προβλήματα έχουν να κάνουν με συστημικές δυσκολίες και αν δεν λυθεί αυτό δεν μπορούμε να περιμένουμε πραγματικά βελτιώσεις. Θα έρθω σε αυτό λίγο αργότερα. Πρώτα απ' όλα πάντως επιτρέψτε μου να σας αναφέρω κάπως τις απλοποίησεις που έχουν ήδη εισαχθεί στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και ποιες από αυτές βοήθησαν πραγματικά να έχουμε κάποια βελτίωση. Θα έρθω πρώτα στην διευκόλυνση της ενία καταχώρησης σε νέα ηλεκτρονικής φύσεως διοικητικά μέσα και τους ελέγχους που οι απαιτήσει για τους ελέγχους αυτούς έχουν μειωθεί. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι έχει διευκολυνθεί το θέμα των, της από τις τράπεζες και ο συντονιστικός ρόλος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει επίσης απλοποιηθεί. Υπάρχουν βέβαια και άλλες απλοποίησεις για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο που ίσως να μην είναι και τόσο ευπρόσδεκτες. Δεν έχουν λειτουργήσει πάντως όπως περιμέναμε, αν μη τι άλλο. Ε, πιστεύω, η Επιτροπή μάλλον πιστεύει ότι η καταποκοπή ποσά, ή άλλα έξοδα, σταθερά ας πούμε έξοδα, αποτελούν απλοποίηση του συστήματος. Αναμφίβολα, μεγάλη απλοποίηση για την Κομισιόν είναι κάτι τέτοιο, αλλά ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει παραπάνω δουλειά για τους δικαιούχους. Και ο λόγος είναι ότι περισσότεροι από αυτούς που συμμετέχουν στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο χρησιμοποιούν πραγματικά έξοδα είναι αλήθεια αυτό για πολλέ επιχειρήσει και μικρέ και μεσέ επιχειρήσει και σίγουρα και για τα πανεπιστήμια. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή τελικά. Σημαίνει ότι αν πάτε τα ξύδι για μία συνάντηση για ένα πρόγραμμα, αγοράζετε ένα αεροπορικό εισιτήριο, πληρώνετε το ξενοδοχείο σα. Η τιμή μπαίνει στου λογαριασμού σαν πραγματικό κόστο για τα έξοδα που κάνατε. Και όταν εσεί πάρετε κατά αποκοπή ε, μια αποζημίωση για τα έξοδα αυτά, τελικά παίρνετε όχι το ποσό το οποίο έχετε δαπανίσει, αλλά κάτι άλλο. Ε, αυτό ε, διορθώνεται με ε, επιπλέον λογιστικές διαδικασίες, κάτι το οποίο περιπλέκει βέβαια το ζήτημα. Χρειάζεται διαφάνεια, να έχουμε τα πλήρη ποσά και αυτό προτιμάμε. Βέβαια, αν υπήρχε μια δυνατότητα ε, σε θελοντική βάση να μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί το σύστημα με καταποκοπήν αποζημίωση, ίσως αυτό να ήταν το καλύτερο. Έπειτα υπάρχει και το θέμα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση. Έχει αποτύχει μέχρι τώρα. Υπάρχουν δύο διαδικασίες πιστοποίησης. Η μία επιτρέπει τους συμβαλόμενους να χρησιμοποιούν τα έξοδα για το προσωπικό εφόσον η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τα έξοδα αυτά τα αποκρίνεται στα κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δυστυχώς τα κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τόσο αυστηρά που τελικά καμία επιχείρηση και κανένας αφορέας δεν μπορεί να αποκριθεί σε αυτά. Κάναμε μία μελέτη σε 30 από τις μεγαλύτερες ε, τέτοιες οργανώσεις στην Ευρώπη και είδαμε ότι το 80% δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε πολλές άλλες περιπτώσεις ε, υπήρχαν ε, μεγάλες αμφιβολίες. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απλοποίηση που θα δημοσιοποιηθεί νομίζω αύριο. Κυκλοφορεί ήδη νομίζω ως σχέδιο και μας λέει ότι 90% των οργανώσεων που χρησιμοποιούν το μέσο κόστος για το προσωπικό δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα κριτήρια τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είχε στόχο την απλοποίηση ε, του κόστους αυτού, αλλά τελικά εμποδίζει τις περισσότερες οργανώσεις να υποφεληθούν από το μέτρο αυτό. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να λυθεί. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η εκτελεστική οργάνωση είχε σαν στόχο την απλοποίηση. Α, όχι. Κάτι δεν πάει καλά με τις διαφάνειες, λέει ο μιλητής. Για να το διορθώσω. Α, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν πρόκειται για απλοποίηση ή όχι, αλλά εγώ δεν βλέπω βελτίωση. Και μάλλον έχουν χειροτερέψει τα πράγματα. Ο χρόνος όμως πιέζει και γι' αυτό δεν θα μπω εδώ σε λεπτομέρειες. Τώρα, κάποια θέματα για τις ε, κοινέ πρωτοβουλίες. Γιατί μετά έχω κι άλλα. Μου ζητήθηκε να πω ποιες είναι οι παρετέρω πλοποιήσεις που θα θέλαμε. Βέβαια διστάζω κάπως γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά δύο προτάσεις θα είχα να κάνω που πιστεύω ότι θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση. Το ένα που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι μια ενιαία ερμηνεία των κανόνων που διέπουν το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και που να ισχύουν για όλες τις γενικές διευθύνσεις, για όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για όλες τις υπηρεσίες. Διότι υπάρχει σύγχυση και δημιουργείται διάκριση σε βάρος ορισμένων όταν ε, διαφορετικές γενικές διευθύνσεις ερμηνεύουν διαφορετικά τον ίδιο κανόνα και ακόμα και οι υπηρεσίε μέσα στην ίδια γενική διεύθυνση μερικέ φορέ ερμηνεύουν διαφορετικά έναν κανόνα. Η λύση για μένα θα ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα σώμα υψηλού επίπεδου που θα φροντίσει να επακούν σε αυτό όλες οι γενικές διευθύνσεις και που θα εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και ερμηνεία των κανόνων που να είναι πράγματα δεσμευτικά για όλες τις υπηρεσίες, για όλους τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ίδιο σώμα θα μπορούσε να λειτουργεί και ως διαιτητικό όργανο κατά κάποιο τρόπο, στο οποίο θα μπορούσαν να προσφύγουν οι δικαιούχοι εφόσον θεωρούν ότι δεν έχει γίνει σωστή ερμηνεία ή σωστή εφαρμογή των κανόνων. Το δεύτερο που θα είχα να προτείνω και που πιστεύω ότι θα απλοποιούσε πολύ τα πράγματα για όλους και για την Επιτροπή και για τους δικαιούχους θα ήταν το κόστος να δηλώνεται σύμφωνα με τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές. Αυτό προβλέπεται για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά στην πράξη εφαρμόζεται δύσκολα, γιατί υπάρχουν και άλλα κριτήρια τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται και δυσκολεύουν αυτή τη δυνατότητα. Αν λοιπόν το κόστος θα μπορούσε να καταγραφεί σύμφωνα με τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές, τότε και εφόσον οι πρακτικές αυτές έχουν εγκριθεί από κάποια εθνική αρχή ελεγκτική, θα γινόταν πιστεύω αυτό. Βέβαια αυτό θα σήμαινε διαφορετικές ε, προδιαγραφές ε, στην κάθε χώρα. Αλλά αυτό νομίζω θα μπορούσαμε να το δεχτούμε. Και μάλιστα θα μπορούσαμε έτσι και να ενθαρρύνουμε κατά κάποιο τρόπο τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών για τις βέλτιστες πρακτικές έρευνας. Και η Επιτροπή θα μπορούσε να έχει συστήματα ελέγχου ώστε οι εθνικές πρακτικές να ανταποκρίνονται σε ορισμένα ελάχιστα κριτήρια. Τώρα θέλω να έρθω λιγάκι στα συστημικά προβλήματα, στο οποίο αναφέρθηκα και πριν, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε κάποιες κάπως περίεργες συνθήκες, θα έλεγα θεσμικούς συστημικούς κινδύνους. Κάτι δεν πήγε καλά και έχει να κάνει με τους κανόνες συμμετοχής. Ο νομοθέτης, δηλαδή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κυρίαρχα καθορίζουν τους κανόνες αυτούς συμμετοχής. Το εκτελεστικό όργανο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, εφαρμόζει τους κανόνες αυτούς και τους εφάρμοσε όπως φανταζόταν ότι ήταν η πρόθεση του νομοθέτη. Το ελεγκτικό συνέδριο όμως ερμήνευσε διαφορετικά τις προθέσεις του νομοθέτη. Και έτσι για πολλά χρόνια επέκρινε την ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κύρια, η κριτική του ελεγκτικού συνεδρίου είναι 10% το πολύ ανεκτό σφάλμα, που κατά τη γνώμη μου και δεν είμαι και ο μόνος, μπορεί να είναι καλό για να ελέγχουμε τις ε, δαπάνες για τις δημόσιες προμήθειες, αλλά δεν είναι το σωστό ποσοστό για τέτοιες δραστηριότητες όπως έχει το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Οι επικρίσεις αυτές λοιπόν επαναλαμβάνονταν κάθε χρόνο και στο Κοινοβούλιο, το οποίο Κοινοβούλιο επίσης επέκρινε την κατάσταση αυτή. Κατέληψε λοιπόν τους κανόνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποφάσισε αυστηρά να τηρεί τους κανόνες. Έτσι, θέλησε όχι μόνο να τους εφαρμόσει για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, αυστηρά τους κανόνες αυτούς, αλλά και για το 6ο, για το παρελθόν δηλαδή, για το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο, με πολύ σοβαρές ε, ε, συνέπειες, διότι έτσι πλήττεται η εμπιστοσύνη των ε, δικαιούχων και αυξάνεται και το διοικητικό κόστο των συμμετοχόντων και υπονομεύεται και η ίδια η πολιτική έρευνας. Μια που η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά γίνεται όλο και λιγότερο ελκυστική. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα κλίμα μεγάλης δυσπιστίας. η διαθεσμική νοτροπία στην Ποέτσι ελέγχου δεν λειτουργεί καλά. Έχει φτάσει σε διαστάσεις που τελικά η απόδοση και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών δεν είναι εφικτή. Ενώ το αντίθετο θέλουμε να πετύχουμε. Τι πρέπει να γίνει, πρέπει να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των συμμετοχόντων στα προγράμματα πλαίσια, το 7ο και τα επόμενα. Ήδη έχουν ξεκινήσει νομικές διαδικασίες, προσφυγές κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από διάφορους δικαιούχους του 7ου προγράμματος πλαισίου. Κάτι λοιπόν πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει και γρήγορα. Διότι η εκστρατεία, ο έλεγχος που κάνει το ελεκτικό συνέδριο έχει προχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα θα αρχίσει να βγάζει ε, εντάλματα για επιστροφή ποσών και θα υπάρξουν σίγουρα και άλλες νομικές διαδικασίες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όταν φτάσουμε εκεί, καταλαβαίνετε ότι η ατμόσφαιρα που ήδη δεν είναι και πολύ καλή, θα έχει γίνει εντελώς δηλητηριώδης. Γι' αυτό λοιπόν όλοι, νομοθέτες, συμμετέχοντες, όλοι πρέπει να συζητήσουν και να καταλήξουν σε μια απόφαση όσον αφορά τη στρατηγική για το 2020. Τα επιχειρήματα που θα σας δώσω, προσέξτε τα πάρα πολύ τώρα παρακαλώ. Όταν ξεκίνησε τους ελέγχους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα πλαίσιο το έκτο, αποφάσισε λοιπόν πολύ αυστηρά να εφαρμόσει τους κανόνες. Αναδρομικά και μονομερός δηλαδή αποφάσισε να αλλάξει την ε, ερμηνεία της όσον αφορά το κόστος. Και έτσι Πρόκειται, σύμφωνα με την Επιτροπή, για παραβίαση των όρων των συμβάσεων. Αλλά πάνω σε αυτό έχουν κάνει δικαιούχοι ε, προσφυγή. Διότι έτσι οι συμμετέχοντες στο έκτο πρόγραμμα πλαίσιο ε, φαίνεται ότι έχουν κάνει παρανομίες και οι πληρωμές που έχουν γίνει δεν είναι σωστές, δεν θα πρέπει να γίνουν. Και εδώ δεν μιλάμε για ελάχιστους ε, αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πλήρωσαν τα ποσά αυτά ε, με κάποιο τρόπο που δεν έπρεπε. Εδώ μιλάμε για μια γενικευμένη στάση από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής προηγουμένως και άρα πρόκειται για τεράστια ποσά. Κατά συνέπεια, οι δικαιούχοι του έκτου προγράμματος οπλαισίου, όχι αλλά συστηματικά ε, βρίσκονται σε λάθος. Είναι δυσανάλογη λοιπόν αυτή η κατάσταση. Θα έπρεπε να γίνει μια ανάλυση για να δούμε τι πλήρωσαν τελικά οι συμβαλόμενοι και να επανεκτιμηθούν τα ποσά για το πρόγραμμα αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να πάρει πίσω ούτε 10 ευρώ για 100 ευρώ που έχει δώσει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι όλη αυτή η διαδικασία κάνει περισσότερη ζημιά στην έρευνα, στην πολιτική έρευνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση παρά καλό στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελώνω με το εξή. Οι περισσότεροι από του συμβαλόμενου κατηγορούνται για σφάλματα τα οποία δεν έκαναν. Είναι απαράδεκτο να τους ζητηθεί να πληρώσουν ε, ποσά για λάθη που έχουν γίνει σε κάποιο άλλο σημείο της αλυσίδας και που δεν έχουν κάνει οι ίδιοι. Θα οδηγήσει αυτό σε θεσμικές διαμάχες. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από όλα τα θεσμικά όργανα να συμφωνήσουν μεταξύ τους να πάυσει κάθε έλεγχος ex post, που αφορά δηλαδή το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση που φαίνεται να έχουν γίνει απάτες ή τεραστίου μεγέθους αμέλειες. Αν το κάνουμε αυτό, θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε καλύτερη διαχείριση του 7ου προγράμματος πλαισίου βάσει των πόρων που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να επικεντρωθούμε λοιπόν στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Άρα λοιπόν προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ελέγχους για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο σε πραγματικό χρόνο. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει ελέγχους επιτόπου. Και έτσι δεν θα υπάρχουν ε, διαφορές όσον αφορά την ερμηνεία των κανόνων και αν υπάρχουν τέτοιες διαφορές θα εντοπίζονται έγκαιρα και θα διορθώνονται. Βέβαια από μόνο του ένα τέτοιο μέτρο δεν φτάνει, γιατί υπάρχει και το θέμα του 2% ανεκτό σφάλμα. Ταυτόχρονα λοιπόν πρέπει να συμφωνήσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, ε, συγγνώμη, το Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο επ' Αν γίνει αυτό και γίνουν συγχρόνω οι έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο και όχι εξπόστ, τότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή του 7ου προγράμματος πλαισίου. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ένωσης Πανεπιστημίων, θα ήθελα να πω δύο λόγια σε ορισμένα σε ορισμένε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων και η δικιά μου χώρα, η Ιταλία, βλέπουμε σημαντικότατε περικοπέ στα πανεπιστήμια. Κάθε μέρα κλείνονται τμήματα των πανεπιστημίων, άρα ε, κλείνει το μέλλον ε, των φοιτητών. Από την άλλη πλευρά ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση των προγραμμάτων κατάρτισης που όμως ε, διαπιστώνουμε ότι τελικά δεν ε, ευωδώνονται και ε, διαπιστώνουμε επίσης και βάσει και των όσων μας είπε και η Όλαφ σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα γιατί το συζητήσαμε χτες γίνονται σημαντικότατες απάτες ε, στα προγράμματα αυτά και επομένως θα πρέπει ε, να δούμε από πολύ κοντά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Κρίστοφερ Χάλ και δίνω το λόγο στον κύριο Τόμα Έστερμαν, ο οποίο είναι προϊστάμενο του τμήματο διακυβέρνηση, αυτονομία και χρηματοδότηση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστήμιων. 15 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας κύριε Έστερμαν. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε ε, και μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα για την ε, πρόταση. Η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ε, εκτιμά ιδιαίτερο την δυνατότητα που της δίδεται να συζητήσει αυτό το θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σας ε, πω πρώτα ποια είναι τα κεντρικά σημεία κλειδιά ε, όσον αφορά την απλούστευση το, της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Εγώ δεν θα αναφερθώ μονάχα στο πρόγραμμα πλαίσιο. Αναφέρομαι ε, και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και στου δικαιούχους αυτή τη ευρύτερης χρηματοδότηση. Να σας πω όμως δύο λόγια πρώτα απ' όλα για την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και να σας πω πώς διαμορφώνομαι άποψη για τα κεντρικά σημεία, μεταξύ των οποίων και η χρηματοδότηση. Είμαστε μια μη κυβερνητική οργάνωση ε, που έχει μέλη 850 μεμονωμένα πανεπιστήμια πολλά ε, τμήματα ε, που ασχολούνται εντονότατα με την έρευνα, όπως ας πούμε την Οξφόρδη. Επίσης με 46 χώρες, έχουμε επίσης περίπου 35 ε, συλλογικά μέλη, Βρετανικά συμβούλια πρέπει να σας πω ότι εκπροσωπούμε τα περισσότερα πανεπιστήμια των χωρών μας. Γι' αυτό λοιπόν ε, πιστεύουμε ότι μπορούμε να εκπροσωπήσουμε αυτόνομα και ανεξάρτητα τον τομέα των πανεπιστημίων. Έχουμε δύο ε, κεντρικά βασικούς πυλώνες ε, που μας βοηθούν να καταρτούμε την άποψή μας. Ε, έχουμε αφενός το Συμβούλιο, ε, το οποίο λαμβάνει γνώση των ερευνητικών προγραμμάτων και εκεί συμμετέχουν πολλοί ερευνητές, εθνικοί φορείς και ερευνητικά κέντρα και ο δεύτερος πυλώνας είναι οι μεμονωμένες έρευνες που κάνουμε σε μεμονωμένα πανεπιστήμια. Εκεί πρέπει να σας πω ότι στο θέμα της απλούστευσης ε, έχουμε κάνει ε, πολλές ε, μελέτες, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ για να δούμε πώς είναι δυνατόν να υπάρξει απλούστευση στα θέματα της πλήρους κοστολόγησης των προγραμμάτων αυτών και έχουμε και ένα πρόγραμμα που τρέχει τώρα, το οποίο λέγεται EUDIS ε, και το οποίο αναφέρεται ακριβώς στη διαφοροποίηση ε, των ε, χρηματοδοτήσεων. Έχουμε ποσοτικά στοιχεία από 200 και πλέον πανεπιστήμια, από 30 και πλέον χώρες έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι τα οχήματα ε, που θα μας οθήσουν προς το μέλλον, ενώ ταυτοχρόνως ε, να δούμε και ποια, ποιες είναι οι τροχοπέδες που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε ας πούμε μέλος ένα πανεπιστήμιο ε, στο οποίο αυτή τη στιγμή τρέχουν, ένα μεγάλο ε, πανεπιστήμιο και ερευνητικό κέντρο, αυτή τη στιγμή τρέχουν περίπου 600 ερευνητικά προγράμματα. Καταλαβαίνετε πόσο προσφυλές είναι για μας το θέμα της απλούστευσης. Κεντρικά σημεία λοιπόν της απλούστευσης. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Είναι πάρα πολύ, σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικό ε, να μιλήσουμε για όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Είναι θέμα αρχής. Το δεύτερο ε, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μία ισορροπημένη και αναλογικά ε, σωστή διαδικασία κοστολόγησης και απόδοσης δαπανών. Τρίτον, η απλούστευση θα πρέπει να αφορά ολόκληρη τη διαδικασία από την εφαρμογή μέχρι την αναφορά και τον ε, ε, λογιστικό έλεγχο. Έγιναν κάποιες ε, βελτιώσεις, αναφέρθηκε ο προηγούμενος ομιλητής σε ορισμένες από αυτές τις νέες μεθόδους, αλλά παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγάλος βαθμός βελτίωσης και απλούστευσης. Θα χωρίσω το υπόλοιπο του, της ομιλίας μου σε τρία θέματα το πρώτο θέμα το οποίο θα ε, αφορά στους κανονισμούς και τι πρέπει να αλλάξει με τους κανονισμούς, δεύτερον στην εφαρμογή και θα τελειώσω με κάποιες λύσεις, δηλαδή κάποια βήματα που μπορούν να ληφθούν στο μέλλον έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Όσον αφορά τους ε, κανονισμούς, το μεγάλο πρόβλημα είναι η πολυπλοκότητα και η πολυμορφία των ε, κανονισμών. Ε, σας είπα και προηγουμένως ότι υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα τα οποία δουλεύουν με ε, πολλούς ε, τρόπους χρηματοδότησης από τα Life and Learning ε, προγράμματα, από διάφορα προγράμματα. Επομένως, η, όταν η εφαρμογή είναι διαφορετική, όταν ο τρόπος απόδοσης είναι διαφορετικός, αυτό σημαίνει ότι περιπλέκεται ιδιαίτερος η η κατάσταση. Επομένως, αυτή η πολυμορφία των κανονισμών ε, θα πρέπει να ειδωθεί λίγο από πιο κοντά όσον αφορά την χρηματοδότηση. Επίσης, είδαμε διαφορετικούς κανόνες ε, διαφορετικό ε, οικονομικό πλαίσιο αλλαγή των κανόνων για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο και επομένως ε, είναι εξαιρετικά σημαντική η απλούστευση αυτών των ε, διαδικασιών. Δεύτερον, υπάρχουν προβλήματα ερμηνείας τα οποία προκύπτουν και από την διαφορετική ορολογία που προκύπτει με τη σειρά της από τα διαφορετικά κανονιστικά και ρυθμιστικά πλαίσια. Επομένως, θα πρέπει να ξαναδούμε την ορολογία η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί, να επιλεγεί αυστηρά και βεβαίως θα πρέπει όσον αφορά την ορολογία να αφαιρεθούν όλα, ε, όλες οι ορολογίες οι οποίες είναι ασαφείς, καθώς επίσης και όλες οι, ε, ε, όλες οι νομοθεσίες, αν θέλετε, ή όλα τα ρυθμιστικά, κανονιστικά πλαίσια, τα οποία το ένα έρχεται σε αντίθεση με το άλλο. Και ξέρετε, έχουμε, αντιμετωπίζουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, δηλαδή ότι ενώ έχει ξεκινήσει μία διαδικασία ε, ε, αλλάζουν ε, οι κανονισμοί και αυτό προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, εμείς θέλουμε το σύνολο των κανόνων να είναι συγκεκριμένο και γνωστό ήδη από την αρχή του προγράμματος. Και αυτό ελπίζω να ισχύσει για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Αναφέρθηκα ήδη στην, ε, ε, στις πολλαπλές μεθόδους και πρέπει να πω ότι τη στιγμή που έχουμε πάρα, πολύ διαφορετικούς, πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού και πάρα πολλούς τρόπους ταυτοποίησης δραστηριοτήτων, ε, στόχους ε, κόστους, στόχους ε, οχημάτων, στόχους βάσης, αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση. Χρειαζόμαστε ένα κοινό λογιστικό σύστημα, κάποιες πρακτικές, λογιστικές πρακτικές που δεν είναι απαραίτητα, απαραίτητο να είναι ακριβώς ίδιες με αυτές που χρησιμοποιεί ο ιδιωτικός τομέας αλλά και ο δημόσιος τομέας θα πρέπει οπωσδήποτε να ενοποιήσει λίγο τις ε, ε, μεθόδους και εν πάση περιπτώσει δεν είναι δυνατόν σε όλα τα τεχνολογικά ιδρύματα ή σε όλα τα ερευνητικά κέντρα να εφαρμοστούν απαράλλακτα οι ίδιοι κανόνες. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια δυνατότητα ε, διαφοροποίησης. Επίσης να σας πω ότι να σας πω ότι τα πανεπιστήμια είναι ιδιαίτερα περίπλοκα ιδρύματα και επομένως ε, λαμβάνοντας υπόψη και το τι συμβαίνει και στα αντίστοιχα ιδρύματα του Καναδά ή των Ηνωμένων Πολιτειών όταν μιλάμε για έρευνα θα πρέπει να δούμε και ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Όσον αφορά την απόδοση των δαπανών πρέπει να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι απόδοσης και αναφοράς. Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι βασικές λογιστικές αρχές να μπορέσουν θεωρητικά να εφαρμοστούν και εδώ. Και βεβαίως πάντα θεωρητικά αυτές οι ε, λογιστικές μέθοδοι κατά κανόνα επιτρέπουν μια διαφοροποίηση. Τελευταίο σημείο όσον αφορά τους κανονισμούς. Ε, θα ήθελα να αναφέρω εδώ σαν τελευταίο σημείο την ε, οικονομική αηφορία. Αυτή τη στιγμή έχουμε σαφέστατη μείωση των δημοσίων δαπανών ε, για την, ε, για την ανώτατη εκπαίδευση και για την ε, έρευνα ιδιαίτερος. Ο προϋπολογισμός για την ανώτατη παιδεία ε, μειώνεται παντού και επομένως δεν καλύπτεται το κόστος των δραστηριοτήτων. Επομένως ε, βλέπουμε ότι ήδη έχουμε ένα χάσμα ε, χρηματοδοτικό το οποίο θα διευρυνθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον και επομένως θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το βήμα της χρηματοδότησης του πλήρους κόστους της ε, έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά θα έχουμε την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε δραστηριότητες έρευνας πάρα πολύ σημαντικές. Όσον αφορά την εφαρμογή, έρχομαι στο δεύτερο σκέλος της ε, παρουσίασής μου, εδώ θα ήθελα να απομονώσουμε τέσσερα σημεία. Το κύριο πρόβλημα είναι η ερμηνεία που δίνεται στους κανονισμούς. Επομένως, πρέπει να έχουμε κάποιες ε, ε, αρχές ε, οι οποίες θα μας οδηγούν και βεβαίως αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές να μην μπορούν να την χάνουν διαφορετικών ερμηνεών. Και βεβαίως θα πρέπει όλη αυτή η διαδικασία να βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Αλλά πώς θα καθοριστεί αυτή η εμπιστοσύνη. Ε, τα πανεπιστήμια θεωρούν μείζονο σημασία στην συνέχιση του διαλόγου έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και βεβαίως καλύτερη κατανόηση της ε, περίπλοκης αποστολής που έχουν τα ε, πανεπιστήμια. Γιατί το πανεπιστήμιο ασχολείται και με τη διδασκαλία και με την έρευνα αλλά έχει και ευθύνες απέναντι στην κοινωνία. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύστημα το οποίο μπορεί να είναι περίπλοκο και στην διαχείρισή του. Και ακόμα και αν κάποιο χρηματοδοτεί μονάχα μία δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει το σύνολο της αποστολής ε, του Πανεπιστημίου. θα πρέπει να βρούμε επίσης βέλτιστες πρακτικές. Ας πούμε, στο Ηνωμένο ε, Βασίλειο ε, υπάρχει μία διαδικασία η οποία έχει οδηγήσει στον έλεγχο, στον, στην, ε, στον έλεγχο του πλήρους κόστους ε, του Πανεπιστημίου και θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει ένα λαμπρό παράδειγμα εφαρμογής ε, κανόνων. Το τελευταίο σημείο που ήθελα να θίξω, ήδη το έθιξε ο προηγούμενος ομιλητής, είναι η πιστοποίηση. Ε, ε η πιστοποίηση είναι ε, πολύ καλή, αλλά παρόλα αυτά και εδώ η απλούστευση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει κανείς να έχει μία συνολική έποψη του ε, συστήματος βάσει των αρχών που ανέφερα και προηγουμένως. Και εδώ πάλι εισέρχεται το θέμα των, ε, της ε, καθαρότητας των κανόνων. Πρέπει το κανονιστικό πλαίσιο να είναι σαφές έτσι ώστε και να είναι κατανοητή και η αποστολή του Πανεπιστημίου έτσι ώστε όλα να πάνε καλά. Ο, τελειώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σε πέντε σημεία τα οποία μπορεί να θεωρηθούν λύσεις ή τα επόμενα βήματα. Πρώτον, θα πρέπει να υπάρξει αναγνώριση της τεράστιας διαφοροποίησης της ανάπτυξης των ε, συστημάτων κοστολόγησης. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα, διαφορετικές ταχύτητες στην ε, ε, ανάπτυξη και τον, του κόστους ε, και στην εξέλιξη του κόστους και δεν είναι δυνατόν να μην το δέχεται αυτό κανείς. Θα πρέπει αντιθέτως να στηριχτεί το σύστημα του, της απόδοσης του πλήρους κόστους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή σαν Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ε, κάνουμε μία έρευνα όσον αφορά το 7ο πρόγραμμα ε, πλαίσιο για να προσπαθήσουμε να, να, δούμε προς τα πού πηγαίνει ε, το κόστος. Αυτό είναι ουσιώδες για μας και μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο πιλότο, οδηγό. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνει προσεκτική ανάλυση του τρόπου εφαρμογής των ε, ισχυών των ε, κανόνων και να δούμε πώς εφαρμόζονται στα διάφορα πανεπιστήμια. και να ε, ε, οριστεί και ένα φόρουμ των εμπλεκομένων ε, και ενδιαφερομένων μερών έτσι ώστε να μπορέσουν να εργαστούν πάνω σε συγκεκριμένα στοιχεία της απλούστευσης θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος, θα πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι ε, και να συζητούν τα θέματα. Εμείς σαν Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ε, είμαστε απολύτως διαθέσιμοι να δώσουμε ε, την πραγματογνωμοσύνη μας κατά αυτή την έννοια. Τέταρτο σημείο, θα πρέπει να διαρευνήσουμε την δυνατότητα να βγάλουμε την χρηματοδότηση της έρευνας από την γενικότερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. θα πρέπει να δούμε ενδεχομένως έναν τρόπο να απομονώνουμε και την ε, ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου έρευνα. Τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω σαν λύση είναι η δημιουργία μιας ομάδας η οποία θα παρακολουθεί την πρόοδο και την εφαρμογή των ε, κανόνων. Πιστεύομαι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια ομάδα η οποία βάσει του ελέγχου θα απομονώνει αμέσως τα προβλήματα έτσι ώστε όσο γίνεται πιο γρήγορα να μπορεί να τα ε, λύνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. και θα δώσω τώρα στο λόγο στον κύριο Έρικ Σούλτς, εκτελεστικό διευθυντή της Αρτέμιδος, που θα μας ε, παρουσιάσει την ε, κοινή τεχνολογική ε, πρωτοβουλία του, της, της ομάδας Άρτεμις. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πρώτα όλες και όλους για την πρόσκλησή σας, αλλά ομολογώ ότι έχω ένα πρόβλημα. Οι πρώτοι ομιλητές σήμερα είπαν ότι έχουν πολύ ε, σημαντικότερα πράγματα να συζητήσουν από τα JTIs, δηλαδή τις ε, Joint Technology Initiatives. Εγώ για αυτά θα σας μιλήσω όμως, θα σας εξηγήσω δηλαδή ποια α, θέματα αντιμετωπίζουμε για τις, ε, για τις κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες. Αυτές οι JTIs είναι ένα νέο όργανο μέσα στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου 7 κατ' εφαρμογή το άρθρο 171 τώρα έχει γίνει το 187 της νέας συνθήκης. Πρώτα θα ήθελα να διευκρινίσω ότι υπάρχουν πέντε ε, τέτοιες κοινέ τεχνολογικέ πρωτοβουλίες που δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα περίπου, αλλά αυτές είναι δύο τύπων. Τρεις που είναι μια συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και κομισιών μόνο, η EMI Clean Sky και το FCH. Η χρηματοδότηση εδώ προέρχεται μοναχά αποκλειστικά από την Κομισιόν. Υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη συμβολή της βιομηχανίας από ό,τι στα συνήθη ε, μοντέλα του ε, FP7 αλλά ο, ο τρόπος χρηματοδότησης είναι ο παραδοσιακός του FP7. Τα άλλα δύο, Artemis και ENIAC, έχουν άλλο μοντέλο. Είναι δηλαδή η βιομηχανία, είναι η Κομισιόν, αλλά είναι και οι χώρες που χρηματοδοτούν τις ερευνητικές Υπάρχει λοιπόν συγχρηματοδότηση της Κομισιόν και των χωρών μελών. Να διευκρινίσω κάτι εδώ για τη σημερινή συζήτηση. Εγώ δεν είμαι ακριβώς ε, απολύπτης τέτοιων χρηματοδοτήσεων, είμαι περισσότερο διαμεσολαβητής. Ε, δηλαδή φροντίζω τα χρήματα που έρχονται από την Κομισιόν να πάνε στα διάφορα ερευνητικά ιδρύματα κλπ. Αυτά τα δύο μοντέλα λοιπόν Artemis και ENIAC. Το πρώτο είναι για ενταγμένα ε, συστήματα υπολογισμού και το δεύτερο είναι για άλλα μέτρα. Ε, τώρα, εάν εξετάσετε για παράδειγμα το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιείται σήμερα και που είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιούσατε πριν από τρία χρόνια. Ο ηλεκτρονικός σας υπολογιστής είναι διαφορετικός από αυτό που χρησιμοποιήσατε παλαιότερα. Αν πάρετε το αεροπλάνο, όταν πετούν τα αεροπλάνα βέβαια. Τα αεροπλάνα ήδη είναι και αυτά διαφορετικά, τα αυτοκίνητα είναι διαφορετικά και όλα αυτά βέβαια είναι επειδή έχει γίνει συνδυασμός μικροηλεκτρονικής και ενταγμένων ε, συστημάτων, ενταγμένης ευφυΐας μέσα στα νέα συστήματα. Embedded ε, δηλαδή technology. Όλα αυτά έχουν μεγάλες απαιτήσεις τεχνολογικές. Η αξιοπιστία η διαθεσιμότητα 24 ώρες την, ε, το 24ωρο και 7 ώρες την ημέρα. Άρα λοιπόν ασφάλεια απέναντι σε ατυχήματα αλλά και απέναντι σε ε, εγκληματικές πράξεις όλα αυτά είναι οι μεγάλες τεχνολογικές απαιτήσεις για τα συστήματα του αύριο. Γι' αυτό το λόγο και εδώ και καιρό, από το 2004 δηλαδή, η βιομηχανία μαζί με την Κομισιόν ξεκίνησε το πρόγραμμα Artemis ως μια πλατφόρμα τεχνολογική δημιουργήθηκε μια ατζέντα στρατηγική για ολόκληρη, ε, για ολόκληρη τον πλανήτη συμμορφόμενη με τις απαιτήσεις της ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ξεκίνησε η πρωτοβουλία αυτή από την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εγώ είχα το προνόμιο τότε να συμπροεδρεύω τη ομάδα εργασία η οποία ε, έκανε την, έφτιαξε την ατζέντα αυτή. Οι πυλώνες αυτού του ναού, αν θέλετε έτσι, και που ισχύουν, εξακολουθούν και υπάρχουν σήμερα είναι τα όργανα που προωθούν την ε, έρευνα στην Ευρώπη. Αριστερά έχετε τα παραδοσιακά του προγράμματος πλαισίου 7. Δεξιά έχετε τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα που υπάρχουν στο περιφερειακό και στο εθνικό επίπεδο Στη μέση έχετε τους δύο αυτούς πυλώνες που βλέπετε. Το ένα είναι το Εύρυκα, γιορέκα, και το άλλο είναι αυτή η κοινή ε, πρωτοβουλία, ε, joint undertaking, η οποία ε, προχωρεί πλέον σε ένα downstream, ένα στα, στα κατάντη δηλαδή, πιο κοντά στο προϊόν, το τελικό προϊόν επομένως. Έχουμε λοιπόν τώρα στην επόμενη διαφάνεια όλα αυτά τα οποία συνεργάζονται. Αριστερά έχετε την Αρτεμισία, στην περίπτωση του Άρτεμις δηλαδή, που είναι ένωση βιομηχανιών που δημιουργήθηκε για να δημιουργηθούν με τη σειρά τους οι JTI, οι κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες. Και βλέπετε διάφορων ειδών ε, μέλη, μεγάλες επιχειρήσεις, μικρές και μέσες επιχειρήσεις, καθώς και ερευνητικά ιδρύματα. Υπάρχει το steering board και το προεδρείο. είχα το προνόμιο να είμαι από τους πέντε ε, ιδρυτές πατέρες της Αρτεμισίας που ιδρύθηκε στο, στις αρχές του 2007 για να προετοιμάσει το έδαφος για τη δημιουργία των JTIs. Δεξιά έχετε τις ε, δημόσιες αρχές. Θα δείτε ότι έχετε τις χώρες μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κομισιόν που είναι που διαθέτουν δηλαδή τη χρηματοδότηση για τις ε, αυτές, ε, για το κοινό αυτό εγχείρημα που λέγεται ε, Artemis. Έχετε στο μέσον λοιπόν την Artemis, έχετε το Governing Board, έχετε τον εκτελεστικό διευθυντή που έχει ένα μικρό γραφείο. Όταν ήμουν μέλος στην Αρτεμισία, εμείς η βιομηχανία είπαμε ότι το νέο αυτό όργανο θα πρέπει η διοίκησή του να είναι ε, να, να, βασίζεται σε μια δομή αποτελεσματική και λιτή. Βέβαια χρειάζεται να συμμορφωθούμε με ορισμένου κανόνες. Θα σας ε, πω όμως και ποιες είναι οι αντιφάσεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο δηλώσεις μου. Στη μέση έχετε την ε, Επιτροπή Βιομηχανίας και Έρευνας που αντιπροσωπεί, που αντιπροσωπεί την, μάλλον τη βιομηχανία και κάνει τις προτάσεις στο Συμβούλιο και από την άλλη μεριά οτιδήποτε έχει σχέση με στόχους χρηματοδότησης, χρηματοδότηση των διαφόρων project, είναι ευθύνη του Public Authorities Board, του Συμβουλίου των Δημοσίων Αρχών. Εγώ προσπαθώ να επιτύχω την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων πλευρών και λειτουργεί μέχρι τώρα καλά. Δεν έχει όμως το εύρος, το μέγεθος που είχε προβλεφθεί αρχικά η συνεργασία αυτή ακόμα. Είπα ότι αρχίσαμε αυτά. Η Artemis ξεκίνησε με management της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί το άρθρο 16 του κανονισμού του Συμβουλίου προβλέπει ότι μέχρι ότου να υπάρξει ε, εκτελεστικός διευθυντής και να υπάρχει και αυτονομία του Joint Undertaking, η Κομισιόν αναλαμβάνει την ευθύνη της διαχείρισης αυτού του Joint Undertaking. Ανέλαβα τα καθήκοντά μου λοιπόν ε, πέρσι το Σεπτέμβριο και τότε έμαθα όλους τους κανόνες που επιβάλλονται σε κοινοτικό όργανο. Όταν ήμουν από την πλευρά της βιομηχανίας είχαμε πει ότι θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι ε, λιτός, ε, ευκίνητος, μικρός, λίγοι εμπειρογνώμονες, μια ομάδα ίσως 10-12 προσώπων, όχι περισσότερο. Στην πραγματικότητα μέχρι τώρα είμαστε όντως 10. Και εάν πάρω την αναλογία ε, γραμματέων για παράδειγμα ανά πρόσωπα που εργάζονται στην Κομισιόν και στην, τα τη βιομηχανία, η διαφορά είναι τεράστια. Δική μου ευθύνη είναι να προσπαθήσω να κρατηθώ όσο γίνεται περισσότερο στα, στις προδιαγραφές της βιομηχανίας. Τώρα, ανακάλυψα ότι με μια μικρή ομάδα 10 μελών ήμουν υποχρεωμένος να καλύψω όλα αυτά, να έχω data protection officer. Ε, επίσης ε, ε, άλλον αξιωματούχο ο οποίος να ασχολείται με την ασφάλεια, με την ασφάλεια της πληροφορικής, external profile manager. Να χρησιμοποιήσω και τη δυνατότητα, είχα και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω το ABAC, Accrual Based Accounting System θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω το σύστημα αυτό. Αν δεν το χρησιμοποιήσω δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις προδιαγραφές. Υπάρχουν και άλλοι agents, initiating, validating, authorizing και ούτω καθεξής. Τα κάναμε όλα αυτά, όπως άρχισα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, την 1η Σεπτεμβρίου και στις 26 Οκτωβρίου εξασφαλίσαμε την αυτονομία. Εγκρίθηκε η αυτονομία μας. Τελειώσαμε? Όχι. Γιατί Έχω συναντηθεί με πολλούς μου ζήτησαν να βάλω έναν full-time internal auditor, ένα οικονομικό ελεγκτή ο οποίος θα είναι πλήρους απασχόλησης. Αυτά είναι ανοησίες. Χρειάζομαι staff committee, σημαίνει ε, επιτροπή προσωπικού, ανάλογη με αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που μας ζητούν να κάνουμε δηλαδή είναι να αντιγράψουμε σε μικρή κλίμακα, σε, 10, σε κλίμακα 10 ανθρώπων, όλη την δομή της Επιτροπής, η οποία βεβαίως έχει χιλιάδες ε, άτομα προσωπικό. Το ελεγκτικό συνέδριο, σε ένα από τα προ, προκατακτικά του σχόλια, μου ζητάει, για παράδειγμα, ο υπεύθυνο ε, ε τεχνολογίας πληροφορικής να είναι να υπάρχει τέτοιος, αλλά δεν έχει νόημα να έχω τέτοιον για 10 πρόσωπα αυστηρή εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις όλων των αρχών του Four Eyes Principle. Δηλαδή να υπάρχει και ένας δεύτερος ελεγκτής. Εμείς είπαμε, αλλά κάναμε ένα λάθος για το θέμα, για να διευκολυνθούμε δηλαδή, αποφασίσαμε να ανοίξουμε δύο λογαριασμούς για να δεχόμαστε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τη βιομηχανία, από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών. Έχουμε λοιπόν δύο λογαριασμούς όπου ε, δεχόμαστε χρήματα και ένα λογαριασμό για να πληρώνουμε. Έχω όμως μόνο έναν accounting officer. Τη στιγμή που μας ζήτησαν και προσπαθήσαμε να κάνουμε μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό υποδοχής στο λογαριασμό αποστολής, θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει αν είχαμε ανοίξει μονάχα ένα λογαριασμό. Η Γενική Διεύθυνση Προπολογισμών της Κομισιόν μου τα μπλοκάρισε όλα και πέρασα δύο μέρες προσπαθώντας να διαπραγματευτώ να μου επιτρέψουν να κάνω μια εξαίρεση και έδωσα ειδική υπόσχεση να παρακολουθώ, για, μόνο και μόνο για να μπορέσω να μεταφέρω χρήματα από το ένα λογαριασμό στον άλλο. Μας έχουν φορτώσει λοιπόν αρχές όπου τελικά είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε περισσότερο τις διαδικασίες παρά την ουσία. Όμως εγώ δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσω σε μια τέτοια εξέλιξη όσο θα έχω τη δυνατότητα να διευθύνω την ε, διαδικασία αυτή και ίσως χρειαστεί να επανέλθω εδώ ενώπιόν σας γιατί ίσως να χρειαστεί να σας ζητήσω απαλλαγή για την ε, χρήση του προϋπολογισμού. Ίσως λοιπόν σε ένα χρόνο από τώρα να χρειαστεί να επανέλθω ενώπιόν σας. Αυτά που ήθελα να πω και νομίζω ότι είναι σημαντικό το μήνυμα αυτό. Εσείς συζητείτε ενδεχόμενες αλλαγές τώρα του χρηματοδοτικού κανονισμού. Σημαντικό. Υπάρχουν και οι κανονισμοί του προσωπικού και αυτοί είναι σημαντικοί. Αλλά δεν αποτελούν αυτά παραμοναχά το πρώτο βήμα της διαδικασίας. Έχετε μετά τους κανόνες εφαρμογής, όπου πολλοί στο περιβάλλον αυτό εδώ, στις Βρυξέλλες εννοώ, κάνουν τα πράγματα ακόμα πιο περίπλοκα. Οι κανόνες εφαρμογής φορτώνουν περιπλοκότητα ε, στην όλη διαδικασία. Και δεν φτάνει καν αυτό, γιατί έχει και το, υπάρχει και το τρίτο βήμα, αυτή η κουλτούρα, ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται οι κανόνες εφαρμογής. Υπάρχει λοιπόν ένα τρίτο στρώμα περιπλοκότητας το οποίο προστίθεται. Η δική μου προειδοποίηση είναι η εξή. Ας αλλάξουμε λοιπόν το χρηματοδοτικό προϋπολογισμό όπου αυτό είναι εφικτό και απαραίτητο. Ας προσπαθήσουμε ωστόσο να απλοποιήσουμε τους κανόνες εφαρμογής και ας προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κουλτούρα, αυτή την οτροπία Ήδη στην ιστοσελίδα μας έχουμε βάλει γιατί είναι σημαντική η έκθεση αυτή. Υπάρχει η έκθεση Σέρπα, όπου προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τι ακριβώς έχει γίνει για αυτές τις πρώτες πέντε JTI. Ποια πράγματα μπορούν να βελτιωθούν και τι αναμένουμε για τις μελλοντικέ ε, εκείνες αυτές τεχνολογικές πρωτοβουλίες. Η έκθεση αυτή, όπως είπα, είναι σημαντική υπάρχουν πολύ σημαντικές συστάσεις που περιλαμβάνονται στο τέλος της εκθέσεως. Και εδώ περιλαμβάνω δύο στην διαφάνειά μου. 1.1. Ναι, υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα τον ένα τέτοιος οργανισμός ευρωπαϊκό όργανο και να ε, σέβεται τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αλλά χρειάζεται αναθεωρημένος κανονισμός. Και όταν λέω αναθεωρημένος εννοώ σοβαρά αναθεωρημένος. Εμείς στην Άρτεμις θεωρούμε ότι χρειάζεται να αλλάχθουν περισσότερα πράγματα, να δοθεί περισσότερη ελευθερία, να γίνουν τα πράγματα πιο απλά. Δεύτερη, η σύσταση που διαλαμβάνω εδώ, η 2.3, ε, να θεσπιστούν συγκεκριμένες και ξεκάθαρες απαιτήσει για τις εκθέσεις που υποβάλλουμε και αναφορές. Το ίδιο και για τις διαδικασίες οικονομικών ελέγχων. Όταν έχετε ένα μικρό ε, σώμα 12-13 ανθρώπων. Γιατί χρειάζεστε τέτοιες απαιτήσει για τους οικονομικού ελέγχου όπως όταν έχετε ένα μηχανισμό χιλιάδων υπαλλήλων. Στην περίπτωση της Artemis και ENIAC, από την πλευρά της Κομισιόν, είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα που μπορεί να έχει κανένας. Όταν παίρνω εγώ χρήματα από την Κομισιόν και τα διανέμω στους τελικούς απολύπτες, Ο ρόλος αυτός είναι σημαντικός. Για να δώσω, δίνοντας ένα ευρώ από τα χρήματα αυτά, παράγεται έργο αξίας 6-7 ευρώ, διότι δίνει η Κομισιόν ένα ευρώ, δίνουν και οι χώρες μέλη το, ε, το δικό τους ποσοστό και πολλαπλασιάζονται τα χρήματα κατά 6 και 7 φορές από αυτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι λοιπόν εργαζόμαστε από κοινού. Είναι αποτελεσματικός ο τρόπος αυτός, είναι αποδοτικός από την πλευρά, από τη σκοπιά δηλαδή τη Κομισιόν. Ας προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε τι διαδικασίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σούλτσου και θα δώσω τώρα τον λόγο στον δόκτωρα Πατρίες Μπέκχολτ, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Technopolis Group, ο οποίος θα μας μιλήσει για την αξιολόγηση των ερευνητικών πολιτικών και προγραμμάτων. 15 λεπτά κύριε Μπέκχολτ έχετε στη διάθεσή σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτέ, κύριε και κύριοι, σα ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε εδώ σήμερα. Μου ζητήσατε να σα μιλήσω για την ε, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του 7ου προγράμματο πλαισίου από πλευρά τη αξιολόγηση. Δεν θα μπω λοιπόν σε λεπτομέρειε όσον αφορά το δημοσιονομικό κανονισμό, την απλοποίησή του κτλ. Αλλά θα πω τι πρέπει να κάνουμε για να ξέρουμε κατά πόσο η χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη είναι όντως αποδοτική και αποτελεσματική. Πρώτα απ' όλα να σας πω ποιοι είμαστε. Ίσως πρέπει να σας εξηγήσω γιατί βρίσκομαι εδώ. Είμαι μέλος της ομάδας Τεχνόπολης που είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός αξιολόγησης χρηματοδότησης για την έρευνα στην Ευρώπη. Έχουμε συμμετάσχει σε πολλές αξιολογήσεις ε, προγραμμάτων και του 6ου και του 7ου προγράμματος πλαισίου. Ε, επίσης βοηθάμε το ελεγκτικό συνέδριο με ειδικέ εκθέσεις όσον αφορά την αξιολόγηση τη έρευνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έχουμε εκπονήσει πολλές αξιολογήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν τα προγράμματα πλαίσιο στα κράτη-μέλη. Έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο στο θέμα της απλοποίησης. Μιλάμε λοιπόν από την οπτική γωνία που είναι ότι βλέπουμε τα προγράμματα πλαίσιο τι λύσανε, τι, σε τι έχουν βοηθήσει. Τώρα, όλοι λένε ο δικός μου τομέας είναι ιδιαίτερος, άρα χρειάζομαι ειδική μεταχείριση. Εδώ έχω να σας πω ότι η έρευνα πράγματι δεν είναι κάτι εύκολο να αξιολογηθεί, η αποτελεσματικότητά της δηλαδή. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε στο μέλλον προκειμένου να μπορούμε να αξιολογήσουμε την έρευνα και ο οικονομικός έλεγχος να ανταποκρίνεται στην έρευνα. Η έρευνα λοιπόν όντως είναι κάτι ιδιαίτερο γιατί εξορισμού είναι κάτι αβέβαιο. Είναι ένα εγχείρημα που ελοχεύει πολλούς κινδύνους. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Αν λοιπόν ζητήσουμε τους συμμετέχοντες σε ένα πρόγραμμα πλαίσιο να μειώσουν τους κινδύνους αυτούς και να κάνουν προτάσεις για έρευνα που δεν ελοχεύει κινδύνους, ε, καταλαβαίνετε ότι θα διηγηθούμε σε ελάχιστες καινοτομίε. Ενώ από την άλλη μεριά χρειάζεται ο κίνδυνος για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποια όρια και να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μεγάλα επιτεύγματα. Άρα λοιπόν εξ ορισμού είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τα αποτελέσματα της έρευνας και εκ των προτέρων να πούμε ότι θα έχουμε μια έρευνα που θα είναι αποτελεσματική, γιατί δεν υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο τι ο κάθε φορολογούμενος θέλει, τα χρήματα που θα δώσει ας πούμε στην έρευνα και το αποτέλεσμα που θα έχουμε από την έρευνα αυτή. Δεν υπάρχει άμεση σχέση, γιατί παρεμβαίνουν πάρα πολλοί παράγοντες. Η κοινωνία θέλει βέβαια την καινοτομία, οι επιχειρήσεις επίσης αλλά δεν είναι εύκολο από τις προσδοκίες που έχει κανείς στην αρχή να ξέρουμε ότι θα έχουμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Μπορεί να έχετε 100 προγράμματα, αλλά άμα κάνετε την αξιολόγηση θα διαπιστώσετε ότι τελικά μικρά προγράμματα, λίγα προγράμματα είναι εκείνα τα οποία είναι πολύ επιτυχημένα και που έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Ενώ πολλά άλλα θα έχουν ελάχιστα αποτελέσματα και δεν θα, έχουν, δεν θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας, στις αρχικές. Άρα λοιπόν ως φορολογούμενος όταν χρηματοδοτείς δεν ξέρεις τι αποτέλεσμα θα έχεις. Υπάρχουν και πολλές μεθοδολογικές δυσκολίες, δεν θα μπω εδώ σε λεπτομέρειες. Πάντως κάτι σημαντικό είναι ότι είναι το θέμα του χρόνου. Αν σήμερα ξεκινήσεις την έρευνα, τα αποτελέσματα θα τα έχει σε 5, σε 10 χρόνια. Έχουμε τέτοια παραδείγματα προγραμμάτων ε, πλαίσιο με χρηματοδότηση τη δεκαετία του 70 από τις επιχειρήσεις και που καταλήγουν μετά από 10-15 χρόνια σε αποτελέσματα. Και μην ξεχνάμε ότι εξαρτάται και από κοινωνικούς παράγοντες, παράγοντες πολιτικής. Δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, η κοινωνία που επωφελείται. Υπάρχουν θέματα όπως είναι η ασφάλεια τροφίμων που μπορεί να επωφεληθεί. Αναπτύσσονται καλύτερες πολιτικές μετά από ένα πρόγραμμα πλαίσιο συχνά. Άρα λοιπόν όλους αυτούς τους παράγοντες πρέπει να τους λάβουμε υπόψη μας αν θέλουμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα. Από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα, τι βλέπουμε. Ότι συχνά με ένα πρόγραμμα πλαίσιο δεν μπορούμε να το απομονώσουμε από το σύνολο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο οδήγησε σε αυτά τα αποτελέσματα, γιατί ένα πρόγραμμα πλαίσιο είναι το κομμάτι ενός παζλ μόνο, που μπαίνει μέσα σε γενικότερο πλαίσιο, στο οποίο συμμετέχουν και τα πανεπιστήμια, οι επιχειρήσεις, με τι δικέ του έρευνε. Άρα λοιπόν τα αποτελέσματα οφείλονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, μέρος μόνο του οποίου είναι ένα πρόγραμμα πλαίσιο. Κάτι άλλο περίεργο με την έρευνα είναι ότι πρέπει να δεχτούμε ότι με αυτά τα προγράμματα που ελοχεύουν κινδύνους μπορεί να έχουμε μια αποτυχία. Αλλά μια αποτυχία δεν σημαίνει ότι χάνονται τα χρήματα. Γιατί μπορεί να οδηγηθούμε σε αποτυχία όσον αφορά του σκοπού του προγράμματος, από την άλλη μεριά όμως έχουμε κέρδη γιατί οι ερευνητές, η βιομηχανία μαθαίνει πράγματα που για παράδειγμα να μην επενδύει. Προς ποια κατεύθυνση δεν πρέπει να πάει. Άρα λοιπόν μπορεί να υπάρχει ο παράγοντας κινδύνου στην έρευνα, αλλά υπάρχει πάντα κάποιο κέρδος. Ένα ευρώ που εντό αγωγικών χάνεται σαν χρήμα, μπορεί να έχει οδηγήσει σε κάποιο άλλο κέρδος γιατί ξέρουμε αν μη τι άλλο ότι από εκεί και πέρα πρέπει να πάρουμε μια άλλη κατεύθυνση. Και αυτό είναι χρήσιμο. Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα πλαίσιο έπειτα σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ένας από τον άλλον. Από τις αξιολογήσεις μας όμως έχουμε διαπιστώσει ότι το διοικητικό βάρος είναι μεγάλο και οδηγεί πολλούς υποψήφιους να μην προχωράνε. Όπως είπαν και άλλοι ομιλητές πριν από μένα, υπάρχει θέμα αξιοπιστίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν είναι μόνο ενοχλητικό το ότι πρέπει να τηρείς όλους τους κανόνες, είναι θέμα αξιοπιστίας. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολλές οργανώσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους και δεν θέλουν να συμμετέχουν σε προγράμματα πλαίσιο γι' αυτό. Άλλοι πριν από μένα τα πάνε αυτά. Απλοποίηση λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει απλοποίηση. Γιατί βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Πρέπει να μπορούμε να προσελκύσουμε και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Να θέλουν να συμμετέχουν. Βλέπουμε επίσης ότι πολλά πανεπιστήμια δεν αναλαμβάνουν συντονιστικό ρόλο. Χάνουμε λοιπόν πολλούς υποψήφιους. Η προσπάθεια που γίνεται σε ένα πρόγραμμα για δικητικούς λόγους, για να μπορούν υπεύθυνοι να λογοδοτούν, όλα αυτά έχουν βαρύνει πολύ τη διαδικασία. Αν απλοποιηθούν, θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε καλύτερα στις καθαρά ερευνητικέ δραστηριότητες. Είναι πολύ δύσκολο για πολλές οργανώσεις να επενδύσουν ξέροντας ότι έχουν πολλές πιθανότητες να κερδίσουν κάτι. Άρα λοιπόν το κυριότερο είναι η απλοποίηση. Μια απλή αίτηση στην αρχή σε ένα πρώτο στάδιο και μετά σε ένα δεύτερο στάδιο να περνάμε σε κάτι πιο περίπλοκο. Αν ε, υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα με δύο φάσεις, δύο στάδια, θα προσελκύσουμε νέους υποψήφιους. Έπειτα, πολλές φορές υπάρχουν νέα μέσα, εισάγονται νέα μέσα και κάθε νέο μέσο που εισάγεται, χρηματοδότησης για παράδειγμα, συνοδεύεται και από νέους κανόνες. Αυτό είναι ένα και τέλος οι δημοσιονομικοί κανονισμοί αποτελούν για πολλούς ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Πολλοί το λένε ότι βαραίνουν υπερβολικά το εγχείρημα της έρευνας. Τώρα, η ερευνητική κοινότητα γνωρίζει πολύ καλά ότι πρέπει να λογοδοτήσει για τα χρήματα τα οποία παίρνει. Μου ζητήσατε να μιλήσω για την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση λοιπόν σίγουρα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέσο για να μπορούν οι υπεύθυνοι να λογοδοτούν. Σήμερα όμως βλέπουμε από τα συστήματα ελέγχου ότι η ισορροπία έχει αλλάξει. Ότι κοιτάμε πολύ περισσότερο το οικονομικό σκέλος, το διοικητικό σκέλος και όχι να κοιτάμε την έρευνα αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ένα μεγάλο αποτέλεσμα, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αναλάβουμε τον κίνδυνο. Και έτσι ο έλεγχος γίνεται κυρίως για το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα, πού πάνε τα χρήματα και πολύ λιγότερο στο περιεχόμενο της έρευνας. Υπάρχουν καλά συστήματα ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αξιολογηθεί το περιεχόμενο της έρευνας. Αν οι υποσχέσεις έχουν οδηγήσει σε κάποια αποτελέσματα. Αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολύ καλύτερα αυτά τα συστήματα. Πάλι έρχομαι στο θέμα της ισορροπίας που σας είπα και πριν, ανάμεσα στον οικονομικό έλεγχο και τον έλεγχο του περιεχομένου της έρευνας. Γίνονται αξιολογήσεις, υπάρχουν οι τρόποι. Το ερώτημα είναι πού θέλουμε να προσανατολίζεται ο έλεγχος. Στο οικονομικό σκέλος ή στο περιεχόμενο. Θα ήταν μεγάλη βελτίωση πιστεύω αν επικεντρωνόμαστε πολύ περισσότερο στο περιεχόμενο λοιπόν και όχι στα αποτελέσματα αυτά καθ' αυτά. Πάντα υπάρχει ένας βέβαια μικρός κίνδυνος όταν πούμε ε, μετρήστε το αποτέλεσμα. Μα άμα θέλουμε να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα, να μετρήσουμε το αποτέλεσμα, πρέπει να ξέρουμε τι αποτέλεσμα περιμένουμε. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα το προκαθορίζουμε από την αρχή της έρευνας, από την αρχή της διαδικασίας. Αυτό όμως δεν είναι σωστό, είναι ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε από πριν να ξέρουμε. Αυτό που συμβαίνει συχνά είναι ότι μετράμε πράγματα που δεν θα πρέπει να μετράμε. Ας πούμε δημοσιεύσεις, ε, παραθέσεις ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Όμως η διπλωματα τεχνιας ομως η αποτελεσματικοτητα της έρευνας είναι κάτι πολύ ευρύτερο από το να κάθεται κανείς και να μετράει τις δημοσιεύσεις. Άρα λοιπόν τα συστήματα ελέγχου δεν πρέπει να περιορίζονται στα πράγματα τα μετρήσιμα, αυτά που μπορούμε να μετρήσουμε, όπως είναι οι δημοσίευσεις για παράδειγμα, ένα σύστημα ελέγχου σίγουρα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το παράγοντα κίνδυνο. Πρέπει να λάβει υπόψη και το γεγονός ότι ε, τα πράγματα αλλάζουν, η τεχνολογία εξελίσσεται. Όταν αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν και τα ερευνητικά προγράμματα και το περιεχόμενό τους. Υπάρχει ήδη, όπως σας είπα, ένα σύστημα ε, μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης και εκθέσεων. Εγώ δεν λέω να χρησιμοποιήσουμε νέα μέσα αξιολόγησης, αλλά τα ήδη υπάρχοντα να τα χρησιμοποιούμε καλύτερα. Τέλος. Το τρέχον σύστημα αξιολόγησης θα μπορούσε να εξυπηρετήσει καλύτερα ε, το πρόγραμμα πλαίσιο, εφόσον βρεθεί καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στον οικονομικό έλεγχο και τον έλεγχο της έρευνας, του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων της έρευνας. Και αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα εφόσον πηγάζει μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή είναι πολύ καλά εξοπλισμένη με συστήματα αξιολόγησης, κυρίως αν το συγκρίνουμε αυτό με το τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Άρα δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο. Μια καλή ισορροπία χρειάζεται για να δώσουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία στα προγράμματά μας. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτό τελειώνω. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μπέκχολτ. Έχουμε τώρα 40 λεπτά στη διάθεσή μας για συζήτηση με ερωτήσεις των βουλευτών και απαντήσεις των εισηγητών. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Μπασιτής. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, nebuvau nusiteikęs pradėti tokios sudėtingos temos, bet e, ką šiandieną mes išgirdom, aš manau, kad e, Υπάρχει ένα πρόβλημα. Όλα αυτά που ακούσαμε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βεβαίως ε, είναι σημαντικό το γεγονός ότι ε, για θέματα χρηματοδότησης ερεύνας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε πολλές επικρίσεις. Και δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που έχω πει ε, ξανά και αυτά που ακούσαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, αναδύθηκαν από την συζήτηση πολλά ενδιαφέροντα και επίγοντα ε, ζητήματα. Οι ομιλητές είπαν ότι η εφαρμογή του έκτου προγράμματος πλαισίου δημιούργησε πολλά προβλήματα στη διαχείριση του συστήματος. Πρέπει να σας πω ότι εγώ είχα πολλές επαφές με προσώπους της Λιθουανικής Πανεπιστημιακής ε, ε, Κοινότητας και και εκείνοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να αλλάξει η στάση μας. Η τελευταία ομιλήτρια ε, από τις κάτω χώρες αναφέρθηκε στο γεγονός ότι και αποτυχημένα εντό εισαγωγικών ε, ερευνητικά προγράμματα μπορεί να έχουν πάρα πολύ θετικό ε, αποτέλεσμα τελικά. Επομένως, ε, μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Επίσης, ε, συμφωνώ ότι έφτασε πλέον η στιγμή να αλλάξει η στάση μας. Δεν είναι δυνατόν να αξιολογούμε μονάχα το κόστος. Θα πρέπει να αναφερόμαστε και στο περιεχόμενο της έρευνας, γιατί μην ξεχνούμε ότι η έρευνα είναι ένας τομέας εξαιρετικά περίπλοκος και επομένως ε, θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τις ε, κατευθυντήριες ε, αρχές μας και να μελετούμε και το περιεχόμενο. Λοιπόν, έχουμε και κάποιες πρακτικές προτάσεις πλέον, οι οποίες μας οδηγούν στην αλλαγή της στρατηγικής μας. Βεβαίως ε, οι μεγαλύτερες χώρες και οι παλαιότερες χώρες ιστορικά έχουν ε, το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης ε, και επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό ιδρυμάτων που δέχονται τη χρηματοδότηση. Άρα πολιτικά πολιτικά, ε, με πολιτικούς όρους θα πρέπει να, να αλλάξει και η στάση μας όσον αφορά την συμμετοχή των χωρών και των πανεπιστημίων γιατί οι νέες και οι μικρότερες χώρες έχουν μικρότερη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα ή σε παλαιά ερευνητικά προγράμματα. Όσον αφορά τώρα την χρηματοδότηση της έρευνας, συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη ή δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μονάχα ε, το, υψηλό περιεχόμενο ενό ερευνητικού ενός προγράμματος ε, έτσι ώστε και απλούστερα προγράμματα να χρηματοδοτούνται. Νομίζω ότι ε, μετά την συνθήκη της Λισαβόνας ε, το Κοινοβούλιο έχει μεγαλύτερο ρόλο στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και επομένως ελπίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε και εφαρμόζοντας τις δερμοδιότητές μας θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα ερευνητικά προγράμματα στο μέλλον τα επιτεύγματα ε, στον επιστημονικό τομέα είναι ε, πάρα πολύ σημαντικά και βεβαίως αποτελούν και κίνητρο για μας να συμμετάσχουμε σε μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα. E, και για τα μελλοντικά λοιπόν προγράμματα ε, πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξουν αυτές οι αρχές. Έχουμε διαθέσιμα για το μελλοντικό ε, ε, πλαίσιο, πρόγραμμα πλαίσιο 126 ε, εκατομμύρια για τα ειδικά ερευνητικά προγράμματα και νομίζω ότι θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους ερευνητέ μας να δουλέψουν σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σοντή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε βεβαίως ε, για την οργάνωση ε, της ε, ακρόασης στο πρώτο μέρος της οποίας ακούσαμε την άποψη των δικαιούχων και βεβαίως περιμένουμε με αγωνία και το δεύτερο τμήμα. Πρώτον, νομίζω ότι η Επιτροπή, η Επιτροπή Βιομηχανίας είναι αυτή η οποία θα πρέπει να ασχοληθεί με το περιεχόμενο και όπως έλεγε και ο στρατηγός Δεγκόλ ε, χρειαζόμαστε ερευνητές αλλά χρειαζόμαστε ε, και αυτούς που θα βρίσκουν πράγματα, όχι μόνο αυτούς που θα ερευνούν. Άρα είναι το περιεχόμενο σημαντικό αλλά και η έκβαση είναι εξίσου σημαντική είναι γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα πλαίσιο προβληματικών διαδικασιών και διεργασιών. Ε, υπάρχουν ένα σωρό ε, υπάλληλοι οι οποίοι χώνουν τη μύτη τους παντού, ακόμα και εκεί που δεν τους αφορά τίποτα. Υπάρχει πολλαπλότητα ανθρώπων, τομέων, διαδικασιών και επομένως τη στιγμή που θα διαπραγματευτούμε τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, ε, τη στιγμή που θέλουμε η έρευνα να γίνεται περισσότερο σε ενωσιακό επίπεδο, θα πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα, αυτή η πολυφωνία. Και τα προβλήματα αυτά στην ουσία δεν είναι και τόσο σοβαρά. Στην ουσία ποια είναι τα θέματα τα οποία μας υπέβαλαν ε, οι δικαιούχοι. Έχουμε συμβάσεις έργου και συμβάσεις επιδότησης ε, οι οποίες ε, ε, κλείνονται βάσει καταποκοπήν εξόδων ενώ έχουμε μετά τον εκ οικονομικό έλεγχο ο οποίος λέει ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτήν την ανάλυση εξόδων. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ συγκεκριμένο το οποίο μπορούμε να βρούμε, στο οποίο μπορούμε να βρούμε λύση. Και τελειώνοντα να πω το εξή. Πρώτον, ο καθένα θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Είπε κάποιο ότι παρεμβαίνοντα ότι χρειάζεται διοργανική συμφωνία μεταξύ ε, ε Κομισιών Συμβουλίου και Ελεγκτικού Συνεδρίου. Α μην βάλουμε ε, το Ελεγκτικό Συνέδριο παντού. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι, ε, για μία, είναι εκεί και ο ρόλο του είναι για μία διασφάλιση του συνόλου των ε, διεργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται να μπαίνει παντού. Και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά αδόκιμο να βάλουμε το ελεγκτικό συνέδριο από την αρχή. Και πιστεύω ότι το ζήτημα θα πρέπει να λυθεί ανάμεσα στους δικαιούχους, την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε το παρελθόν. Αυτό είναι κεφαλαιόδου σημασία. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε ε, διάφορους ερευνητικού οργανισμούς με την δαμόκλεια σπάθη να κρέμεται πάνω τα κεφάλια τους. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το παρελθόν οι δικαιούχοι με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς οικονομικούς ελέγχους ε, καμιά φορά δίνουν αντιφατικούς, ε, αντιφατικά αποτελέσματα σε σχέση με αυτά της ε, Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστεί το παρελθόν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όσον αφορά το μέλλον θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού έτσι ώστε να δούμε μαζί με τους οργανισμούς έρευνας και τους εκπροσώπους τους, να δούμε, λέω, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια σωστή απλούστευση, έτσι ώστε να μην ξαναβρούμε μπροστά μας τα ίδια προβλήματα και άρα να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Η κυρία Γκρέσλε. Τώρα ας μην συζητούμε αν το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Ε, στην έρευνα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω όλες τις ομιλίες διότι είμαι και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών και εκεί συζητούν το θέμα της, υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων. Πάντως το θέμα της έρευνας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο έλεγχος του προϋπολογισμού δεν αποτελεί τμήμα του προβλήματος αλλά αποτελεί τμήμα της λύσεως το τονίζω αυτό. Εδώ και χρόνια έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα και στο πρόγραμμα πλαίσιο 6 και στο πρόγραμμα πλαίσιο 7. Ήμασταν και από τους λίγους εκείνους που προτείναμε λύσεις. Είμαστε λοιπόν με την πλευρά των καλών. Αυτό είναι πρώτα το μήνυμα που θέλω να αποστείλω στην Κομισιόν, άλλωστε έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη, ότι δηλαδή οι θέσεις που έχει λάβει το Κοινοβούλιο και υπάρχουν σχετικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη και άκουσα και ότι ο κύριος Κρίστοφερ Χάλ τοποθετήθηκε με παρόμοιο τρόπο. Επίσης θεωρώ ότι όλοι μπορούμε να διδαχθούμε κάτι από την κατάσταση αυτή. Το πρώτο δίδαγμα πρέπει να είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ομοιομορφία αλλά και αποδοχή των διαφορών. Για παράδειγμα στην ορολογία. Δυσχεραίνουμε το έργο μας. Διαρκώς επινοούνται νέα μοντέλα συνεργασίας. Εγώ όμω έχω ανάγκη να μου τα εξηγήσετε αυτά τα πράγματα εν τέλει. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ούτε εμεί οι ίδιοι πλέον έχουμε εικόνα, έχουμε επισκόπηση. Να εγγύψετε, και ζητώ από την Κομισιόν, στα πραγματικά προβλήματα. Έχω κάνει προσπάθεια να, να περιλάβω τα σημεία κριτικής που έχετε υποβάλει εσεί στην εργασία μας. Υπάρχει μια μελέτη που δείχνει καθαρά ότι το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κανόνες οι οποίοι έρχονται και επιβάλλονται πάνω σε, νέους, σε παλαιότερους κανόνες και έτσι έχει, έχουμε χάσει πλέον πραγματικά την επισκόπηση. θα πρέπει να καθίσει κάποιο να εξετάσει αν όντω εφαρμόζονται όλοι αυτοί οι κανόνε. Γιατί αλλιώ τι νόημα έχει να θεσπίζονται διαρκώ και νέοι. Πρέπει να συζητήσουμε και μέσα στα πλαίσια της συζήτηση του δημοσιονομικού κανονισμού το ζήτημα του ανεκτού κινδύνου που πρέπει να περιλάβει την λύση όλων των μεγάλων προβλημάτων. Πάντως, προσοχή. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι πρώτα πρέπει να εξετάσουμε τους κανόνες τους οποίους έχουμε ήδη θεσπίσει. Να τους εξετάσουμε, να τους απλοποιήσουμε εκεί όπου πρέπει να απλοποιηθούν, αντί να λέμε ότι καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία δεν μας αρέσουν και τα πετάμε τα συμπεράσματα στο καλάθι των αχρήστων. Δεν γίνεται έτσι. Η συζήτηση για τον ανεκτό κίνδυνο εν τέλει αποτελεί μια διέξοδο για να μείνουν τα πράγματα όπως είναι. Πρέπει να τηρήσουμε τα υπεσχημένα κυρίως εκεί όπου είπαμε για απλοποίηση των κανόνων. Όμως πρέπει να δεχτούμε και την διαφορά των διαφόρων συστημάτων απόδοσης λογαριασμών. Διερωτώμε με, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν διεθνείς λογιστικοί κανόνες και διεθνείς λογιστικές προδιαγραφές. Πώς λοιπόν δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε ότι αυτοί οι κανόνες θα ισχύουν για όλους. Έτσι γίνεται άλλωστε και στην οικονομία γενικότερα. Εν τέλει, η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι δυσχερής. Διότι χρειάζεται ισότιμη μεταχείριση όλων που υποβάλλουν στους λογαριασμούς. δεν εφαρμόζουμε το ίδιο, πρόγραμμα, το ίδιο σύστημα συγγνώμη, ελέγχων που εφαρμόζουμε για παράδειγμα στη Γεωργία, όπου γίνονται έλεγχοι ε, του, της τάξης του 5%, τη του 5%. Ε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί το ίδιο και εδώ. Εμεί πάντω συμπαρατασσόμαστε μαζί σας και απευθύνομαι στους ομιλητέ μας εδώ, γιατί θέλουμε να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερε ανάγκες και απαιτήσει των ερευνητών. Βλέπω ότι από το έκτο και μέχρι το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δεν πετύχαμε να βελτιωθεί η συμμετοχή των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Κάπου οφείλεται αυτό. Χρειαζόμαστε λοιπόν καινοτόμε προσεγγίσει. Με λίγα λόγια εν τέλει θέλω πρώτα να σας ευχαριστήσω και για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα των προτάσεών σας που θα δεχθούμε και θέλω το κεφάλαιο της έρευνας στον δημοσιονομικό κανονισμό να διευρυνθεί και να μπορέσουμε εν τέλει με τους κανόνες που έχουμε, του δημοσιονομικού κανονισμού, μετά τους rules of participation. Αυτοί οι rules of participation, οι κανόνες συμμετοχής, να ενταχθούν στον δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτό θα επιτύχει μια σημαντική απλούστευση. Ήδη με την μείωση του αριθμού των κανόνων θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μια σημαντική απλούστευση. Γι' αυτό λοιπόν και είναι καλόδεχτες οι προτάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τόγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την οργάνωση αυτού του, αυτής της ενδιαφέρουσας ακρόασης γιατί πρέπει να πούμε ότι διαπιστώσαμε ε, μια πολύ ε, μεγάλη σαφήνεια ανάλυσης από τους ε, παρεμβαίνοντες, καθώς επίσης και μεγάλη διάθεση να συζητήσουν μαζί μας. Νομίζω, και όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι συνάδελφοι που ακολουθούμε από καιρό, παρακολουθούμε από καιρό το πρόβλημα, το τομέα της έρευνας, ότι συχνά διαπιστώσαμε τα προβλήματα. Και πολύ συχνά Είδαμε καλές ιδέες, ας πούμε, τις τεχνολογικές πλατφόρμες, αλλά αλλά διαπιστώνουμε επίσης ότι με τη σειρά των ετών είτε αυτές οι καλές ιδέες ε, μερικώς μονάχα εφαρμόστηκαν ή απέτυχαν ή ότι από την άλλη πλευρά, ενώ ήταν καλές ιδέες, δεν κατάφεραν να υλοποιηθούν γιατί τα εργαλεία χρηματοδότησης, γιατί η δυνατότητα βοήθειας ή στήριξης ήταν ελλειπή. Ξεκινήσαμε λοιπόν το 2004 με τις ε, τεχνολογικές πλατφόρμες που είχαν ε, πολύ στρατηγικές ε, αναλύσεις διαφόρων πραγματικών μετά περάσαμε στις ε, κοινέ τεχνολογικές ε, ε, πρωτοβουλίες και ήδη τον Οκτώβριο του 2009 είχαμε κάποια αποτελέσματα ελπέστατα και από το 2002 μέχρι το 2009 τελικά άξιζε τον κόπο όλη αυτή η διαδικασία και τελικά να ρωτήσω σαφώς, λειτουργούν οι κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες, λειτουργούν ή όχι, γιατί αν διαπιστώσαμε ότι δεν λειτουργούν, τότε να τι σταματήσουμε, να μην κάνουμε άλλες. Φοβούμε, φοβούμε ότι αυτές ε, οι JTIs, οι οποίες ε, στην ουσία είναι επιχειρήσεις, στις JTIs λοιπόν εμείς αναπαράγουμε την ε, Κομισιόν. Δηλαδή, ίδιος τρόπος λειτουργίας, ίδιος τρόπος ε, ε, υπαλληλικής νοοτροπίας, ίδιος τρόπος διαμόρφωσης υπαλληλικού σχήματος. Δηλαδή, τι, αναπαράγουμε μικρές Κομισιόν. Αλλά τι κάνουν τελικά, έχουν αποτέλεσμα αυτές οι επιχειρηματικές δομές. Έχουν όμως την αυτονομία, δεν ξέρουμε πώς επιλέγουν το προσωπικό τους. Λειτουργούν λοιπόν σαν μονάδες. Είναι δυνατόν όμως να ζητήσουμε από αυτές τις ιδιωτικέ, ας το πούμε επιχειρήσεις να αναπαράγουν τον τρόπο λειτουργία τη Κομισιόν που είναι ένα δημόσιο φορέα. Υπάρχουν ένα σωρό ωραίες ιδέες, ας πούμε με τα κύτταρα υδρογόνου ή ας πούμε έρευνα για φάρμακα. Ε, όλες αυτές οι αναλύσεις είναι πάρα πολύ καλές. Το, το θέμα είναι πώς μπορούμε να περάσουμε από τις αναλύσεις σε αποφάσεις. Ακούσαμε και γνωρίζουμε πολύ συχνά τις δυσκολίες ε, που ε, υπάρχουν και αντιμετωπίζουν ε, τα τεχνολογικά ιδρύματα από τη στιγμή της ανάθεσης μέχρι τον τελικό έλεγχο. Ρωτώ λοιπόν, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων βάσει των οποίων αυτοί που, ενδιαφέρονται, που ενδιαφέρονται αναρωτιούνται γιατί πρέπει να χάσουν ένα σωρό χρόνο έτσι ώστε να υποβάλουν την αίτηση. Ε, εδώ δεν χρειάζεται θαύμα για να γίνουν αλλαγές. Μία απόφαση της ε, Κομισιόν που να λέει να αλλάξουν οι διαδικασίες έτσι ώστε να απλουστευτούν οι διαδικασίες. Ε, συνήθως μας λένε ότι να, το κοινοβούλιο είναι το ε, ο, ο φύλακας ας πούμε ο οποίο γαυγίζει κάθε φορά που λέμε να απλουστεύσουμε τι διαδικασίες γιατί το κοινοβούλιο θέλει διασφαλίσεις κτλ. Εγώ έχω συναντήσει πάρα πολλά τεχνολογικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, ιδιώτες που λένε ναι ναι θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να υποβάλουμε την αίτηση αλλά χρειάζεται μια στίβα χαρτιά και δεν είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Και νομίζω ότι αν δούμε ε, τώρα το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο θα διαπιστώσουμε ότι και η αξιολόγηση κόστους ωφέλους θα πρέπει να γίνει. Εκεί όπου υπάρχει ε, οποιαδήποτε απάτη, οποιαδήποτε έλλειψη, ναι βεβαίως να παρέμβουμε και να παρέμβουμε μάλιστα αποφασιστικά. Αλλά ε, ε, διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν όλες οι διαδικασίες. Ε, δηλαδή να βρούμε έναν άλλο τρόπο, να μην ανοίξει μια απίστευτη, ένας απίστευτος γύρος αντιπαραθέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας ε, ε, συγχαρώ, να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η ιδέα που είχατε για την οργάνωση της ακρόασης και θέλω να κάνω μια ερώτηση και στους τέσσερις ουσιαστικά, γιατί ο καθένας από αυτούς προέρχεται από ένα διαφορετικό χώρο, από μια διαφορετική δομή, που έχει εμπειρία σε τοπικό, σε εθνικό επίπεδο καταρχήν, και άλλοι έρχονται από το Πανεπιστήμιο που έχουν εμπειρία σε διεθνή συνεργασία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω, όλα τα προβλήματα τα οποία θέσατε έχουν να κάνουν μόνο με το γεγονός ότι το επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί μια παραπάνω δυσκολία. Ο εκπρόσωπος της Αρτέμιδος, για παράδειγμα, είπε ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός, οι προδιαγραφές που εφαρμόζεται, το καταστατικό του προσωπικού κλπ. Αναφέρθηκε σε αυτές, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι πρόκειται για κάτι τόσο περίπλοκο ή τόσο δύσκολο τουλάχιστον σε επίπεδο εθνικό ή τοπικό. Ίσως επειδή είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό θέλω να μάθω αν είναι αυτή η διάσταση που δημιουργεί δυσκολία. Χρειαζόμαστε επίσης κάτι πιο ιδιαίτερο. Η τελευταία μιλήτρια νομίζω αναφέρθηκε σε αυτό. Αν είναι ένας δημοσιονομικός κανονισμός ο οποίος εφαρμόζεται σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, για άλλες ανάγκες, θα ήταν αλλιώς. Είναι οι παράγοντες αξιολόγησης που δυσκολεύουν τα πράγματα. Θα ήθελα να μπουν περισσότερο σε βάθος. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η κυρία Τόγια για τις υποψηφιότητες. Εμένα με εξέπληξε πράγματι ότι υπάρχουν πανεπιστήμια που δεν έχουν πια τη διάθεση να συμμετάσχουν. Πρέπει να γίνει λοιπόν αυτή η προσπάθεια ώστε να έχουμε περισσότερες υποψηφιότητες και έτσι να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη επιλογή. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα. Η ε, κυρία Ματουρέλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, καλεσμένους μας για την σαφήνεια των λόγων τους. Ευχαριστώ και σας Πρόεδρε που είχατε την ιδέα να οργανώσουμε αυτή την εξαίρετη ακρόαση. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Συμφωνώ μαζί τους με τα περισσότερα. Ε, επίσης όμως να προσθέσω ότι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι η απλοποίηση είναι στοιχείο κλειδί. Γι' αυτό και χαίρομαι που η Ισπανική Προεδρία έβαλε την απλοποίηση στις προτεραιότητές της. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα σε είπαν οι καλεσμένοι μας. Αλλά υπάρχουν προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν. Οι κανόνες της συμμετοχής, ο δημοσιονομικός κανονισμός είναι πράγματα τα οποία πρέπει να φροντίσουμε να διορθώσουμε στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο γιατί εδώ που έχουμε φτάσει με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο δεν νομίζω ότι έχει νόημα να προσπαθήσουμε τώρα να προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε. Γιατί θέλει πολλή δουλειά, προετοιμασία. Όμως, ακούστηκαν και ζητήματα που πιστεύω ότι με τα σημερινά ρυθμιστικά πλαίσια θα μπορούσαμε να αλλάξουμε. Είμαστε στη μέση του 7ου προγράμματος πλαισίου. Οπότε η ερμηνεία των κανόνων είναι κάτι για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε ε, να βοηθήσει. Το θέμα της επανεισαγωγής των ελέγχων εξάντε αντί να γίνονται μετά. Και σε αυτό αναφέρθηκαν πολλοί. Ή το θέμα του ανεκτού σφάλματος. Είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να διορθωθούν τώρα χωρίς να χρειάζονται τεράστιες ρυθμιστικές αλλαγές. Έτσι θα διευκολυνόταν η κατάσταση όσον αφορά το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Έχω και μια ερώτηση. Το θέμα του συντονισμού ανάμεσα στον εθνικό έλεγχο και στον έλεγχο που γίνεται από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μήπως θα μπορούσε να γίνει κάτι για να βελτιωθεί αυτός ο συντονισμός. Διαπιστώνω ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν μεγάλες διαφορές που έχουν οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα τους ερευνητές. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτού και να μην περιμένουμε το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο για να τα διορθώσουμε όλα. Μερικά πράγματα μπορούμε ήδη να τα κανονίσουμε από τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, πολύ σύντομα, κύριο Σοντή. Ναι, μια και δεν έχουμε παρέμβαση της όλα στο δεύτερο τμήμα, υπάρχει ένα ζήτημα ε, των ε, απατών. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ ε, ευαίσθητο θέμα και επίσης ο ανέτιος πλουτισμός είναι θέματα πολύ σημαντικά. Θέλει κάποιος από τους εισηγητές να απαντήσει στις ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοι βουλευτές. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Prego. Ci sono state diverse domande. Ε, έγιναν διάφορες ερωτήσεις. Ποιος θα απαντήσει πρώτος. Well, I would like to uh, respond to the question. Um, θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση που τέθηκε σχετικά με το εάν αυτού του είδους τα προβλήματα και οι δυσκολίες υπάρχουν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή και σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να πω ότι Έχουμε μεγάλο ποσοστό μαρτυριών από διάφορες χώρες. Βεβαίως στις διάφορες χώρες μεμονωμένα υπάρχει έτσι περιπλοκότητα της ε, ε, της χρηματοδότησης, αλλά κάποια διάμεσα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε γενικές γραμμές είναι πιο περίπλοκα από τα εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης. Επίσης, ε, ότι ε, υπάρχουν ε, διαρκώς από πλευράς ε, των ερευνητικών κέντρων ε, υπάρχει γραμμή κατά κάποιο τρόπο που λέει ότι εάν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα χρηματοδότησης από εθνικά προγράμματα να προτιμήσουν τα εθνικά προγράμματα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ανησυχητικό γεγονός, είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Ελοχεύει ο κίνδυνος ο, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να μην επιτύχει τελικά το στόχο της, να μην φτάσει καν μέχρι τα ερευνητικά κέντρα και τα ερευνητικά προγράμματα. Η συμμετοχή των οργανισμών ε, ε, είναι σημαντικός έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επίσης, το θέμα δεν είναι αν θα υπάρχουν ε, ε, κανόνες εφαρμογής, βεβαίως πρέπει να υπάρχουν. Το ζήτημα είναι αν μέσω των ισχυών των κανόνων εφαρμογής μπορούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την καλύτερη δυνατή χρήση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Επίσης ε, είναι καλό να δούμε, ε, να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις ε, με την έρευνα στην Αυστραλία, στις Ηνωμένε Πολιτείες. Να δούμε δηλαδή με ποιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον βέλτιστο τρόπο την χρηματοδότηση. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να, ε, σε αυτό πρέπει να αποσκοπεί και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δηλαδή να μην βλέπει μεμονωμένα προγράμματα, να έχει σαν υπόβαθρο το γενικότερο ε, πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας. Κάποιος άλλος από τους συγητές, παρακαλώ. Εγώ να απαντήσω στα σχόλια που έκανε η Ιταλίδα βουλευτής για τα JTI. Ξεκινήσαμε το 2004 και χρειάστηκαν Τέσσερα-πέντε χρόνια μέχρι ό,τι τα βάλουμε να λειτουργήσουν. Τώρα όμως λειτουργούν οι κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες. Είναι μια, σαν ένα υπέροχο μοτέρ Φεράρι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι το ρεζερβάρ της βενζίνης πότε είναι μισογεμάτο, πότε είναι μισοάδιο. Θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερα οι χώρες μέλη. Λειτουργεί όμως. Από το πρώτο στο δεύτερο και από το δεύτερο στο τρίτο βήμα και έχω και ένα σχόλιο ακόμη για τον έλεγχο κόστους. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες όπως η Artemis είναι ότι εγώ βασίζομαι στις χώρες μέλη και στην δική τους αποδοχή και απόδειξη πληρωμών, δηλαδή προκαταβολών να προσθέσουν το 16,7% του κόστους, όπως αναγνωρίζεται από τις χώρες μέλη. Σε πλήρη συμμόρφωση των τοπικών κανόνων και τοπικών κανόνων ελέγχων. Ακόμα και στην περίπτωση ε, zero funding contracts ή χωρών που δεν είναι μέλη της Άρτεμις πάλι τότε χρειάζεται να εφαρμόζω τους κανόνες του ε, προγράμματος πλαισίου 7, του 7ου δηλαδή. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Εσείς. Ο Κρίστοφερ Χάλ. Τέθηκε το ερώτημα εάν τα πράγματα είναι καλύτερα στο εθνικό επίπεδο Υπάρχει βέβαια μια ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα σε όλο αυτό. Και ο μέγας όγκος της χρηματοδότησης της έρευνας δαπανάται τέλει σε εθνικό επίπεδο. Στις περισσότερες χώρες θα βρείτε συμφωνημένα ε, λογιστικά πλαίσια που να χρησιμοποιούνται για την κοστολόγηση των διαφόρων προγραμμάτων έρευνας. Δεν θυμούμε τώρα πόσες χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμα πλαίσιο, πάντως ο αριθμός τους είναι μεγάλος και είναι προφανώς δύσκολο να υπάρχει ένα ενίο λογιστικό πλαίσιο το οποίο να είναι ταυτόχρονα συμβατό με πολλά εθνικά πλαίσια. Επομένως αυτό δίνει μια ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα. Όπως είπα και εγώ, αλλά είπε και η κυρία Γκρέση, λέει ότι ίσως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν αυτές, υπάρχουν αυτά τα εθνικά εγκεκριμένα συστήματα, ο κόσμος εργάζεται στη βάση αυτών και γιατί δεν μπορούμε άραγε να δεχθούμε κάποια συστήματα και να τα εφαρμόσουμε και για τους ευρωπαϊκούς σκοπούς μας. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, ορισμένοι μίλησαν για τον δημοσιονομικό κανονισμό, ότι αυτός βρίσκεται στη βάση του προβλήματος. Εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες. Όταν έκανε δημόσια διαβούλευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον δημοσιονομικό κανονισμό, προσπαθήσαμε να αναλύσουμε και τον κανονισμό και τους κανόνες εφαρμογής και ειλικρινά δεν βρήκαμε και πολλά εκεί τα οποία να είναι ιδιαίτερα ευνηδιαστικά. Μα φάνηκαν λογικά τα πράγματα. Αυτό που αποτελεί το πρόβλημα είναι η υπερβολική ερμηνεία των κανόνων αυτών. Και επανέρχομαι σε αυτό που περιέγραψα, ίσως εσφαλμένα, ως μια νοοτροπία ελέγχου διαθεσμική η οποία έχει αναπτυχθεί και η οποία εμποδίζει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε λίγο πιο αποστασιοποιημένα και με λίγο πιο χαλαρό τρόπο και τότε θα βρούμε κάποιες λύσεις. Very shortly on the... Για το θέμα της Ισπανίδας ε, Ευρωβουλευτού που είπε ότι πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο αναθερούμε ε, τα προγράμματα πλαίσιο πιο συστηματικά. Επικεντρωνόμαστε τώρα στο εξή. Κάνουμε τα πράγματα καλά, δαπανώνται τα χρήματα με σωστό τρόπο. Όμως η πραγματική πρόκληση που έχει μπροστά της η Ευρώπη είναι κάνουμε το σωστό, δηλαδή δαπανώμε τα χρήματά μας με τρόπο ο οποίος βοηθάει την έρευνά μας να γίνει περισσότερο καινοτόμος τη βοηθάμε να αντιμετωπίσει κοινωνικά ζητήματα που ζητούν λύση. Τα μέσα αξιολόγησης υπάρχουν για να δώσουμε απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα αυτά καλύτερα, να τα πάρουμε περισσότερο στα σοβαρά, για να δούμε κατά πόσο οι στόχοι αυτοί επιτυχάνονται. Είναι θέμα περισσότερης προσοχής στο περιεχόμενο και όχι τόσο το να δούμε αν τα χρήματα δαπανώνται σωστά ή όχι. Δεν φτάνει αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης. Νέες πρόπτικες προς ένα βελτιωμένο πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην εκπρόσωπο της Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου, την κυρία Μιλάγρο Καντέλα, επικεφαλή Σύμβουλο Επιστημών και Καινοτομίας στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ισπανίας. Παρακαλώ. Θα έχετε 15 λεπτά στη διάθεσή σας. Ε, ε, Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην ακρόαση αυτή. Είναι μια ακρόαση που εμείς θεωρούμε ότι αποτελεί ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο σε όλη την διαδικασία συζήτησης και προβληματισμού για την βελτίωση της συμμετοχής στα ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα καινοτομίας που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας εξηγήσω λίγο ότι η Ισπανική Προεδρία το θέμα αυτό της απλοποίησης, της συμμετοχής στο, στα προγράμματα πλαίσιο και γενικότερα σε όλα τα προγράμματα στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας. Το θέμα αυτό λοιπόν ε, το έχει πάρει η Ισπανική Προεδρία πολύ σοβαρά, επειδή πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μας είπε ότι σκοπεύει τώρα την άνοιξη του 2010 να ετοιμάσει μία ανακοίνωση. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα θεσμικά όργανα για να συνεισφέρουμε και εμείς στη ζήτηση που υπάρχει από πλευράς της επιστημονικής κοινότητας και όλων όσων συμμετέχουν στα προγράμματα πλαίσιο. Η Ισπανική Προεδρία μέχρι τώρα προσπάθησε να βάλει στις ράγες τη συζήτηση και οργάνωσε ένα σεμινάριο τον Φεβρουάριο του 2010 όπου πολλοί από τους συμμετέχοντες στην ακρόαση αυτή ήταν και εκεί οι Εκεί ακούσαμε πολλές ιδέες, πολλές σκέψεις, πολλούς προβληματισμούς και μετά από το σεμινάριο αυτό και βάσει των συμπερασμάτων του ετοιμάζουμε μία πρόταση ώστε το Συμβούλιο Υπουργών στην επόμενη συνεδρίασή του, το Συμβούλιο ανταγωνιστικότητας, δηλαδή τμήμα έρευνα, να υιοθετήσει αποφάσεις για κατευθυντήριες γραμμές, για προσαναλωτισμούς που ίσως δεν ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας, αλλά θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες. Υπάρχει και η πρόταση αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού που θα βοηθήσει και που πιστεύουμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά που εμείς δεν θα πειράξουμε στα δικά μας τα συμπεράσματα. Όπως έλεγα λοιπόν, έχουμε ένα σχέδιο συμπερασμάτων για το Συμβούλιο που συζητιέται αυτή την εποχή στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Εγώ θα σας αναφέρω κάποια από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται εκεί και κάποια από αυτά έχουν ήδη συζητηθεί εδώ, τα ακούσαμε. Στην αρχή σήμερα νωρίς νωρίς δεν μπόρεσα να έρθω εδώ γιατί είχαμε ένα τριμερή διάλογο, βλέπετε, όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που πέτυχε. Και γι' αυτό δεν ήρθα εδώ από την αρχή της ακρόασης. Το σχέδιο συμπερασμάτων για την πολιτική στήριξη, τη στήριξη των Υπουργών στο επόμενο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει με απλοποίηση τις διαδικασίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τις αιτήσει, την αξιολόγηση, την επιλογή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο των ενισχύσεων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. Επίσης πιστεύουμε ότι είναι καλό να δούμε δύο θέματα που δεν φαίνονται κεντρική σημασία για το θέμα που μας ασχολεί εδώ σήμερα, αλλά που εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα είναι προσανατολισμοί για να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε την συμπληρωματική χρήση άλλων μέσων και προγραμμάτων κοινοτική χρηματοδότησης. Πέρα δηλαδή από τα προγράμματα πλαίσιο έχουμε και προγράμματα καινοτομία και ανταγωνιστικότητα και έχουμε και τα διαφορετικά ταμεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σωστά προσανατολίζει ένα μεγάλο μέρος των ε, κονδυλίων από τα διαφροντικά ταμεία στην έρευνα και στην καινοτομία. Και πολλές φορές ακούμε παράπονο ότι είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσει κανείς συμπληρωματικά τις ενισχύσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, ή τρίτον, μιλάμε και για την βελτίωση που θεωρούμε ότι είναι αναγκαία όσον αφορά την ενημέρωση και την διαφάνεια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας. Αναφέρουμε διάφορες αρχές που πρέπει να ισχύουν. Την αρχή της απλοποίησης με λιγότερους κανόνες που να είναι διάφανοι και καλά συμφωνημένοι. Μείωση επίσης των περιπτώσεων όπου χρειάζεται επιπλέον ερμηνεία των κανόνων. Μιλάμε επίσης για την συνοχή των κανόνων, την εναρμόνιση των κανόνων, έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες κάθε φορά που πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Ακόμα και αν μιλάμε για διαφορετικά προγράμματα ή διαφορετικά μέσα χρηματοδότησης. Κάτι άλλο που πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό είναι η σταθερότητα και η νομική βεβαιότητα. Οι κανόνες δηλαδή πρέπει να είναι σταθεροί, να ισχύουν πάντα και η ερμηνεία τους να είναι η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις. Κάτι άλλο που έχουμε ακούσει πολλές φορές και που μας βρίσκει σύμφωνος είναι ότι η χρηματοδότηση πρέπει να επικεντρώνεται στην εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στους ερευνητές θέλω να πω και στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Λαμβάνοντας υπόψη βέβαια ότι πρέπει να γίνεται και έλεγχος του δημοσίου χρήματος. Πρέπει να βρούμε δηλαδή μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην εμπιστοσύνη που θα δείξουμε στους ερευνητές και από την άλλη μεριά στον έλεγχο των δαπανών. Κάτι άλλο που πιστεύουμε σημαντικό και που ίσως να χρειάζεται περισσότερη συζήτηση είναι η χρηματοδότηση η οποία έχει σαν βάση τα αποτελέσματα. Αν βασιστούμε στην αριστεία, υπάρχει ο κίνδυνος ε, για την έρευνα. Πρέπει να υπάρχουν και τα δύο. Κάτι άλλο που ακούστηκε εδώ και που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που συζητάμε για την απλοποίηση είναι η αρχή της ε, συμβατότητας. Δηλαδή να αποφεύγουμε επικαλύψεις όσον αφορά την απόδοση λογαριασμών. Επιμένω εδώ γιατί το έχω ξανακούσει αυτό. Έπειτα πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα. Δηλαδή να σχεδιάζουμε καλά τα μέσα που χρησιμοποιούμε στα διάφορα προγράμματα έτσι ώστε να μπορούμε συμπληρωματικά να χρησιμοποιούμε τις διάφορες ενισχύσεις. Αναφέρουμε και διάφορες προτάσεις στο σχέδιο αυτό συμπερασμάτων που προωθούμε στο Συμβούλιο και που συζητιέται αυτή την εποχή. Και μεταξύ άλλων σας αναφέρω μια πρώτη κατηγορία προτάσεων που έχουν ως στόχο να μειώσουν ε, την ε, περιπλοκότητα των διαδικασιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όντω έχει προτείνει διάφορε διαδικασίε. Μερικέ από αυτέ υποχρεωτικά είναι περίπλοκε, αλλά άλλε μπορούν να μην είναι περίπλοκε. Πιστεύουμε επίση ότι πρέπει να μειωθεί ο αριθμό των μέσων. Τώρα έχουμε πάρα πολλά μέσα χρηματοδότησης στη διάθεσή μας που οδηγούν σε ένα περίπλοκο σύστημα τελικά και που δεν είναι πάντα αναγκαία. Κάτι άλλο που πιστεύουμε ότι είναι ζωτική σημασία είναι να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αξιολόγηση του κόστους βάσει των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και βάσει των ε, προσπαθειών που γίνονται για να επιτευχθούν τα αποτελέσματα αυτά. Πολύ περισσότερο δηλαδή έτσι να κάνουμε την αξιολόγησή μας παρά βάσει του κόστους. Έτσι αποφεύγουμε και πολλές, πολλούς ελέγχους ex post. Τώρα μακροπρόθεσμα πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν και πολλά για να πετύχουμε αυτό που εντοπίζουν διάφορες αξιολογήσεις των προγραμμάτων πλαίσιων εδώ και χρόνια που είναι να βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο στο σχεδιασμό των προγραμμάτων και κυρίως όσον αφορά τους διαγωνισμούς. Η πρότασή μας είναι να γίνονται bottom-up, από κάτω προς τα πάνω, και να αποφεύγονται οι λεπτομέρειες και ενδείξεις που έχουν να κάνουν με το μέγεθος, ή την σύνθεση των επιχειρηματικών ομίλων. Να αποφεύγουμε δηλαδή πολύ συγκεκριμένα θέματα. Πρέπει να είμαστε περισσότερο ανοιχτοί, ώστε η την συνθεση των επιχειρηματικων ομηλων να αποφευγουμε επιστημονική κοινότητα και οι συμμετέχοντες στα προγράμματα πλαίσιο να εκφράζουν τις επιθυμίες τους και τις προτάσεις τους. Ε, μια άλλη ομάδα προτάσεών μας έχει να κάνει με τους προσανατολισμούς σε σχέση με την ε, μείωση της έντασης των ε, ελέγχων. Και αυτό μπορεί να γίνει εφόσον έχουμε περισσότερη εξάντε αξιολόγηση. Θέλουμε οι προσπάθειες απλοποίησης να επικεντρωθούν στην αρχή της διαδικασίας, όταν πρόκειται δηλαδή για τους διαγωνισμούς, για την ε, αξιολόγηση και την επιλογή. Έτσι, η αξιολόγηση πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στα τεχνικά στοιχεία και κάτι που θεωρούμε επίσης σημαντικό είναι η μείωση, θα έλεγα η απάλληψη σχεδόν, της διαδικασίας διαβουλεύσεων είναι μια διαδικασία η οποία καθυστερεί πάρα πολύ. Εμείς πιστεύουμε ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. Και θέλουμε να κάνουμε και μια πρόταση που ίσως βέβαια να ακούγεται δύσκολη, να μην την καταλαβαίνει κανείς εύκολα, να μην μπορεί να τις εφαρμόσει, αλλά η επιλογή εκείνων που αξιολογούν τα προγράμματα. Η επιλογή αυτή πρέπει να ενισχυθεί. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να σκεφτεί να φτιάξει μια επιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων που να βοηθάει στην επιλογή των ε, ανθρώπων που αξιολογούν, που συμμετέχουν στα πάνελ αξιολόγησης στο πρώτο στάδιο επιλογής των προτάσεων. Μια άλλη ομάδα προτάσεών μας είναι προσανατολισμοί που έχουν να κάνουν με την διαλειτουργικότητα, όπως είπα και πριν, να μπορούν συμπληρωματικά να χρησιμοποιούνται οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις Και τέλος έχουμε και μια ομάδα προτάσεων για την πληροφόρηση και την διαφάνεια. Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι με αυτά που είπα μέχρι τώρα έχετε καταλάβει το πνεύμα των προτάσεών μας προς τα κράτη-μέλη προκειμένου να εγκριθούν πολιτικοί προσανατολισμοί από πλευρά των Υπουργών Έρευνα στις 26 Μαΐου στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Κάτι άλλο το έχετε καταλάβει, αλλά θέλω να το ξαναπώ, ότι αυτές είναι προτάσεις της Προεδρίας που ακόμα δεν έχουν στηρίξει ομόφωνα όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι τα τέλη Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας σε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα ακρόαση. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, Κύριε Μιλάκρο Σκαντέλα από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ισπανίας. Τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κλάρα Ντελατόρε, η Διευθύντρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, αξιότιμοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ κύριε Δημαντζίστης για την πρόσκλησή σας. Μου φάνηκαν οι προηγούμενες ομιλίες και παρεμβάσεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και στροφή σκέψη. Είναι και υψηλό, έχουν βάλει υψηλά τον πύχη. Θα έρθω σε ορισμένα θέματα και μετά θα υπάρχει χρόνος για ε, συζήτηση. Είναι προφανές, αλλά θα το επαναλάβω, ότι δεσμευόμαστε ως ε, θεσμικό όργανο υπέρ της απλούστευσης και συμφωνώ με πολλές από τις απόψεις που ακούστηκαν σήμερα το πρωί. Έχει λοιπόν γίνει ε, πρόοδος στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο σχετικά με την ε, απλούστευση όπως είπαν και οι ενδιαφερόμενοι. Παρ' όλα αυτά η πρόσβαση στα προγράμματά μας και η σύνταξη των προτάσεων εξακολουθούν να είναι δύσκολες και ιδιαίτερα να τις αισθάνονται δύσκολες οι νεοεισερχόμενοι. Και το διοικητικό βάρος είναι, εξακολουθεί να θεωρείται πολύ υψηλό με μακρές χρονικές καθυστερήσεις. Η αρχή του 7ου προγράμματος πλαισίου επέφερε και έναν αριθμό απλουστεύσεων, απλοποίησεων που αναφέρθηκαν προηγουμένως και οι οποίες ορισμένες από αυτές έχουν ενταχθεί μέσα στις νομικές διατάξεις του ε, προγράμματος πλαισίου, άλλες έχουν, έχουν μπει στο πεδίο της εφαρμογής. Ορισμένες από αυτές αναφέρθηκαν ήδη, αλλά θα υπενθυμίσω ορισμένες από τις ε, ε, επιτεύξεις του FP7. Για παράδειγμα, καταφέραμε να οργανώσουμε το σύστημα με τέτοιο τρόπο ώστε η εκ των προτέρων έλεγχοι και τα αναθεωρημένα προστατευτικά μέτρα για οικονομικά ασθενέστερους συμμετέχοντες ε, να έχουν μειωθεί. Και αυτό έγινε ιδιαίτερα για να διευκολύνει την πρόσβαση μικρών και μεσών επιχειρήσεων και high-tech startups, αυτούς που ε, ξεκινούν δηλαδή σε υψηλές τεχνολογίες. Σημαντική ε, μείωση λοιπόν στον αριθμό των πιστοποιητικών και των δημοσιονομικών δηλώσεων που είναι απαραίτητο να υποβάλλονται. Μείωση λοιπόν της ε, γραφειοκρατίας και του κόστους. Βάλαμε και την Unique Registration Facility ώστε να αφαιρέσουμε κάποιο από το βάρος ε, να μην είναι υποχρεωμένοι δηλαδή να υποβάλουν τα ίδια έγγραφα ξανά και ξανά μέσα στο σύστημα. Ε, επιφέραμε την εκ των προτέρων πιστοποίηση της μεθοδολογίας λογιστικών ελέγχων αναγνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά πάντως το κόνσεπτ θεωρούμε ότι είχε το δυναμικό να ε, φτάσει σε κάποιες απλουστεύσεις. Έχουμε βελτιώσει, έχουμε ελαφρώσει, ελαφρύνει μάλλον τις απαιτήσει για project reporting και ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσετε ότι έχουμε κάνει κάποια πρόοδο και στην βελτιστοποίηση των ε, ε, μέσων μας ηλεκτρονικής τεχνολογίας, τεχνολογίας της πληροφορικής και βεβαίω και την διάδρασή μας με τους ε, ε, δικαιούχους. Να βελτιώσουμε και τις υπηρεσίες μας προς τους ε, δικαιούχους. Συμφωνούμε βέβαια ότι αυτά δεν αρκούν και ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε περισσότερο. Μια άλλη πτυχή της απλοποίησης είναι ότι έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει στην μείωση των ποσοστών σφάλματος. Και εδώ νομίζω συμφωνούμε όλοι στην παρούσα Επιτροπή και πολλοί από το κοινό. Ένας όμως βαθμός περιπλοκότητας, όπως είπαν και άλλοι προηγουμένως, ένας βαθμός περιπλοκότητας των κανόνων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας είναι αναπόφευκτος, διότι οι κανόνες αυτοί συχνά και πιστεύω συνήθως ε, θεσπίζονται για να επιτύχουν στόχους πολιτικής. Και δεν είναι απλή η πολιτική αυτή που καλούμαστε να εφαρμόσουμε. Άλλη σημαντική πτυχή της απλοποίησης είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην επιδίωξη διαφορετικών στόχων πολιτικής, που μπορεί να είναι και πολιτική στόχοι, και την προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών. Προηγουμένως είπαν κάποιοι ότι είναι απαραίτητο να μειωθούν οι διαθέσιμοι μηχανισμοί. Ίσως να γίνει αυτό με αυτόν τον τρόπο. Λέχθηκε επίσης και συμφωνούμε και εμείς ότι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση απλοποίησης μιας διαρκούς απλοποίησης θα πρέπει να είναι η σταθεροποίηση των υφιστάμενων κανόνων. Οι επαφές με τους ε, απολύπτες, με τους δικαιούχους δηλαδή, και έχουμε κάνει μια δημόσια διαβούλευση εμείς, και πολλοί από τους δικαιούχους μας είπαν ότι η σταθερότητα των κανόνων προτιμάται απέναντι στην αλλαγή προς την κατεύθυνση κάπως απλούστερων κανόνων διότι ε, συμμόρφωση με νέους κανόνες σημαίνει νέες διαδικασίες που και αυτά έχουν ε, βεβαίως ε, κόστος. Πολύ συχνά λοιπόν η εισαγωγή νέων κανόνων, έστω και αν αυτοί οι νέοι κανόνε είναι απλούστεροι, σημαίνει ωστόσο μια νέα πηγή περιπλοκότητα. Σε τις μέρες αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει μια ανακοίνωση προς το Συμβούλιο Υπουργών, προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προ την Επιτροπή Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην οποία ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα απλοποίηση υπό το ισχύον νομικό πλαίσιο, αλλά θα διερευνά και επιλογές για μια βαθύτερη και πιο μακροπρόθεσμη απλοποίηση, κυρίως μέσα στα πλαίσια του ε, προγράμματος πλαισίου 8 αυτή η ανακοίνωση περί απλοποίησης, η οποία θα αναφέρεται σε πολλά από τα θέματα που ακούστηκαν σήμερα και πολλές από τις ενδεχόμενες λύσεις που επίσης ακούστηκαν σήμερα, έχει ως στόχο να ξεκινήσει μια ευρεία διαθεσμική, διοργανική συζήτηση και να επιτρέψει σε εμάς, την Κομισιόν δηλαδή, να αναζητήσουμε νέα κόνσεπτ για τη χρηματοδότηση της έρευνας. Όπως για παράδειγμα την αμφιλεγόμενη, και λέω αμφιλεγόμενη γιατί ακούσαμε ορισμένου ομιλητέ που ήταν αντίθετοι, αμφιλεγόμενη λοιπόν χρήση τον, τη συστηματική, την συστηματική χρήση των flat rates, των καταποκοπήν δηλαδή ποσών και ούτω καθεξής. Η απλοποίηση λοιπόν είναι βασικός στόχος και άλλων πρωτοβουλειών που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ε, είπαμε και μέσα στα πλαίσια της αναθεώρησης των δημοσιονομικών κανονισμών και των κανόνων εφαρμογής τους που αποτελούν το γενικό νομικό πλαίσιο για την διαχείριση της ε, κοινοτικής χρηματοδότησης και βεβαίως και των δαπανών για την έρευνα. Και επομένως η επιτυχής αναθεώρηση θα αποτελέσει ε, βασική προϋπόθεση για περαιτέρω απλοποίηση. Όσοι γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις αυτές στο προσεχές μέλλον. Όπως ελέγχθηκε πάλι από προηγούμενους ομιλητές, μία μείζον πρόοδος στην απλοποίηση απαιτεί μία επανεξισορρόπηση ανάμεσα στην ε, εμπιστοσύνη και στον έλεγχο, στην ανάληψη κινδύνων και στην αποφυγή κινδύνων. Όποια και αν είναι τέλος πάντων αυτή η ισορροπία που θα επιλεγεί, θα πρέπει πάντως να διασφαλίζει την υγιή ε, χρηματοδότηση και την υγιή διαχείριση χρηματοδότησης. Και εδώ θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τον λεγόμενο ανεκτό κίνδυνο. Με όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα αυτά μάλλον είναι ε, στενά διασυνδεδεμένα και αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε θα παρακαλέσω την Επιτροπή σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Στρέφομαι στο ε, λεγόμενο ανεκτό κίνδυνο σφάλματος. Θα καθορίσουμε το κόστος των ελέγχων σε σχέση με το ποσοστό σφαλμάτων που έχουμε ε, ανακαλύψει ότι υπάρχει. Ο ανεκτός λοιπόν κίνδυνος σφάλματος και η απλοποίηση έχουν δύο πτυχές. Από τη μια μεριά υψηλότερο ποσοστό ανεκτού κινδύνου μπορεί να επιτρέψει να απλοποιήσουμε κάπως διαδικασίες αφού θα υπάρχουν λιγότεροι έλεγχοι. Από την άλλη μεριά, ωστόσο, οι απλοποιημένοι κανόνες και διαδικασίες μπορούν από μόνες τους να συμβάλλουν στην μείωση του σφάλματος, του κινδύνου σφάλματος. Ε, υπάρχει λοιπόν ένας, ένα είδος κύκλου που ανανεώνεται. Λοιπόν, συνεχίζεται το έργο αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ήδη ένα προκαταρκτικό συμπέρασμα το οποίο θα ήθελα να σας ε, υποβάλω. Το ελεγκτικό συνέδριο του 2008 ανέφερε ποσοστό σφάλματος στην, στο χώρο της έρευνας περίπου της τάξης του 3% με το παρόν επίπεδο ελέγχων. Τα στατιστικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε καθιστούν σαφές ότι η μείωση σημαντικά του ποσοστού σφάλματος θα σημάνει βεβαίως σημαντική αύξηση του κόστου. Και για να φτάσουμε στο 2%, στο benchmark του 2% κατέτος που ε, ζητεί το ελεγκτικό ε, συνέδριο μπορεί να αποδειχθεί απαγορευτικό από αψη κόστους. Το να συμφωνήσουμε λοιπόν σε ένα ανεκτό ε, κίνδυνο σφάλματος άνω του τρέχοντος 2%, του benchmark του 2%, μιλούμε για τους κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται τώρα και που θα διαρκέσουν για πολλά χρόνια ακόμα, για άνω του 2% λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, αποδίδει καλύτερα την ισορροπία ανάμεσα στο κόστος του ελέγχου και στην περιπλοκότητα των ε, ε, όρων επιλεξιμότητας οι οποίοι προκαλούν το σφάλμα και να υπάρχει ένας δικαιολογημένος κίνδυνος σφάλματος θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφύγει το πρόσθετο κόστος και βάρος των έξτρα ελέγχων. Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με απλούστερους και πιο εύχριστους κανόνες θα γίνει μια ε, θα επιτευχθεί μια νέα ισορροπία ανάμεσα στους ελέγχους και θα επιτρέψει την ανακάλυψη περίπλοκων και οργανωμένων μηχανισμών απάτης, που έχουν σημαντικά βέβαια και βαριά αποτελέσματα. Ορισμένοι μίλησαν για τις κοινοπραξίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εμείς δεχόμαστε ότι υπάρχει ακόμα ανάγκη να γίνει πολλή δουλειά για να βελτιωθεί το συνολικό ε, πλαίσιο για την έρευνα. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσφατη για τις ε, κοινόπραξίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που βέβαια χαρακτηρίζονται από κάποια ε, δυσχέρεια προβλεψιμότητας. Η ανακοίνωση λέει επίσης ότι υπό το φως των πρώτων εμπειριών με τις ε, κοινοπραξίες, με τις κοινέ αυτές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει όλες τις ενδεχόμενες επιλογές για την αναθεώρηση στο μέλλον του νομικού πλαισίου. Και οι πρόσφατες συστάσεις ε, της ομάδας των ΣΕΡΠΑ που ανεφέρθηκαν προηγουμένως θα αποτελέσουν ένα σημαντικό follow-up στην ε, ε, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κοινοπραξίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θεωρούμε αυτές τις κοινοπραξίες ως ξεχωριστά όργανα και θα επιτρέψουμε και, θα, θα, δώσουμε συγκεκριμένες διατάξεις. Θα δοθεί λοιπόν ένα νέο πλαίσιο για τις PPP αυτές που θα περιλαμβάνουν και τις ε, κοινέ τεχνολογικέ πρωτοβουλίε, Θα φροντίσουμε ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν στη βάση ενός βελτιωμένου ε, πλαισίου ελέγχων και διαχείρισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απολύτω δεσμευμένη να κάνει επιτυχία, να καταστήσει επιτυχία το FP7 για τις κοινέ ε, τεχνολογικές πρωτοβουλίες. Μιας και έχω τον λόγο θα ήθελα να έρθω στο γιατί δεν αυξάνουμε τους εκ των προτέρων ελέγχους ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστη εκπλήξη στο τέλος. Ας μην λησμονούμε ότι αυτοί εκ των προτέρων έλεγχοι οδηγούν εν τέλει ε, σε ε, χρονικές καθυστερήσεις για να δοθούν οι χρηματοδοτήσεις. Αλλά πάντως υπάρχει δυνατότητα αυτή. Θέλω να τονίσω επίσης τα όσα λέχθηκαν από κάποιον από τους ομιλητές προηγουμένως, ότι χρηματοδοτούμε δηλαδή μια περίπλοκη πολιτική, αλλά και σε ένα περίπλοκο περιβάλλον. Υπάρχουν περίπου 100 χώρες που συμμετέχουν, 100 χώρες παραλαμβάνω, στις, ε, ε, στο πρόγραμμα πλαίσιο, με διαφορετικούς κανόνες, με διαφορετικά πλαίσια κτλ. Και οι τα περισσότερα από τα project είναι multi-partner, έχουν δηλαδή πολλούς εταίρους από πολλές χώρες. Να λοιπόν γιατί προκύπτει αυτή η περιπλοκότητα. Θα αρκεστώ σε αυτά ε, κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι οι απόψεις μου ε, συνέβαλαν ε, στην εξέλιξη της συζητήσεως και βεβαίως είμαι στην διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερωτήσει έχετε και βεβαίως αν με επιτρέπετε θα ζητήσω και πάλι την υποστηρίξη του Κοινοβουλίου στην προσπάθειά μας αυτή. Ευχαριστούμε πολύ την Διευθύντρια Ντελατόρε και θα δώσουμε το λόγο στο, στο μέλος του Ευρωπαϊκού Ελληνικού Συνεδρίου, κύριο Χάραλντ Νόακ. Uh, structured and um, sophisticated meeting. Χαίρομαι που με προσκαλέσατε σε αυτήν την εξειζητημένη και προχωρημένη συνεδρίαση κατά την οποία γίνεται μια προσπάθεια να συγκεραστούν τα αιτήματα των δικαιούχων με τις απαντήσεις και τις προοπτικές της άλλης πλευράς. Στα δικά μου 15 λεπτά θα κάνω και εγώ λοιπόν τη δικιά μου προσπάθεια. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ασχοληθώ με κάποια από τα θέματα που αναφέρθηκαν στο πρώτο τμήμα, ε, όσον αφορά δηλαδή την άποψη των δικαιούχων. Δεν νομίζω ότι εσφάλω όταν λέω ότι οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ε, της ευρωπαϊκής έρευνας, αλλά δεν είναι δυνατόν να καλύψει και όλα τα συμφέροντα ή ενδιαφέροντά τους. Βεβαίως κατανοώ ότι οι δικαιούχοι έχουν ειδικά συμφέροντα, ειδικά ωφέλη, αλλά ο σκοπός ε, των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι το μεγαλύτερο δυνατό κοινό όφελος. Και βεβαίως ε, οι προσπάθειές μας συνδέονται και με την πολιτική στρατηγική. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό το πρώτο τμήμα της ακρόασης το ζήτημα των εθνικών δαπανών. Παλιότερα Ήμουν ε, μέλος ε, του Γερμανικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και πολλοί λόγος γινόταν για τον έλεγχο ε, και την, την λογιστική ανάλυση των χρηματοδοτήσεων της έρευνας, το σκοπό της έρευνας και πρέπει να σας πω ότι και τότε και στη Γερμανία οι δικαιούχοι είχαν πολλά παράπονα από την κατάσταση που επικρατούσε. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε με κάποιο τρόπο την ε, πρόοδο του ελέγχου των διαδικασιών, κοστολόγησης και ελέγχου. Ε, στην Γερμανία έχουμε δύο επίπεδα ελέγχου. Έχουμε το ομοσπονδιακό και έχουμε και των κρατηδίων. και ενδεχομένως ε, θα πρέπει και εδώ να προβλέψουμε και τον κρατικό έλεγχο, ένα ενδιάμεσο πεδίο. Πιστεύω ότι και το ζήτημα της ευελιξίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και έγινε λόγος και για αυτό το θέμα όσον αφορά το πρόγραμμα Artemis. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή τη στιγμή ε, Υπάρχουν και κάποιες αλλαγές βέβαια γιατί μπαίνουν και νέα μέλη. Έχουμε κάποιες, ε, θα, υπάρξει κάποια αναδιάρθρωση των, ε, του οργανογράμματος. Πάντως, εγώ προσωπικά μαζί με την ελεκτική μου ομάδα ελέγχομαι την ε, Artemis και είναι γεγονός και συμφωνώ με αυτό ότι οι ειδικέ οργανώσεις χρειάζονται ειδικό λογιστικό έλεγχο και το κάνουμε αυτό. Βεβαίως κατανοούμε ότι η βάση θα πρέπει να είναι ο δημοσιονομικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να διευρύνουμε τον ορίζοντά μας με άλλες υποχρεώσεις, να βρούμε κάποιους ειδικούς, κάποιες ειδικές οικονομικές ρυθμίσεις. Και όταν θα κάνουμε την Declaration d'assurance για το Artemis, την πιστοποίηση την τελική δηλαδή δήλωση αξιοπιστίας για το Άρτεμις. Ελπίζω να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και κατά αυτή την έννοια νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε και κάποια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ειδικέ καταστάσεις. Ας έρθουμε τώρα σε αυτά που μας απασχολούν στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης. Και να πω αυτό που είπε ο Αντε Σεντεξιπερί ο οποίος είπε ότι η τελειότητα είναι, έχει επιτευχθεί ε, όχι όταν δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα, αλλά όταν δεν χρειάζεται να αφαιρέσουμε τίποτα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η φράση του Αντουάν Τεσεντεξιουπερί δείχνει ε, ότι θα πρέπει να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις ε, για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και επομένως χρειάζεται ε, συμβατεί και ενιαία ερμηνεία των κανόνων και αυτό ε, μπορεί να επιτευχθεί μονάχα εάν οι κανόνες είναι ε, αρκετά ομοιογενείς. Και νομίζω ότι εκεί έγκυται και η ουσία του προβλήματος. Εμείς δεν ερμηνεύουμε τους κανονισμούς με τρόπο διαφορετικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι σωστό αυτό που ακούστηκε ότι εμείς ερμηνεύουμε ε, τους κανονισμούς διαφορετικά από την Επιτροπή. Όμως, καμιά φορά ε, εμείς διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σφάλματα και το υπογραμμίζω. Σφάλμα, δεν, ε, το σφάλμα δεν συνδυναμή με απάτη και αυτό το υπογραμμίζω. Όμως εμείς στον έλεγχο των κανονιστικών ρυθμίσεων διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν λάθη. Αυτό όμως, δηλαδή το ότι εμείς απομονώνουμε κάποια λάθη, δεν σημαίνει ότι δίνουμε διαφορετική ερμηνεία σαν ελεγκτικό συνέδριο από αυτήν που δίνει η Επιτροπή. <coughs> Αλλά βεβαίως ε, ε, ριζική απλούστευση είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός και εμείς σαν ελεγκτικό συνέδριο έχουμε πει επανειλημμένο ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η απλούστευση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ε, για την έρευνα. Επιτρέψτε μου τώρα να, σας, να αναφερθώ ε, στο, στις εξελίξεις του πρόσφατου πλαισίου. Το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια γι' αυτό. Να σας πω τι έγινε όταν ξεκίνησε αυτή η χιλιετία την οποία διανύουμε τώρα. Τότε είχαμε το ε, επέμπτο πρόγραμμα πλαίσιο και το ελεγκτικό συνέδριο στο, στην ετήσια αναφορά της του 2001, δηλαδή 9 χρόνια πριν, ζήτησε λοιπόν μια ουσιώδη απλούστευση του τρόπου επιστροφής του ε, κόστους για το επερχόμενο τότε έκτο πρόγραμμα πλαίσιο. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο πρότεινε να υπάρχουν τρεις ε, κύριες ε, κατηγορίες ε, κόστους το δηλαδή ε, τα επιπλέον κόστη, το πλήρες κόστος και το καταποκοπήν κόστος να ε, ε, αντικατασταθεί από ένα ενιαίο σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θα μείωνε και τις τρεις προηγούμενες κατηγορίες αυτές των προσωπικών εξόδων, των συντονισμένων εξόδων και των ειδικών εξόδων και με τον τρόπο αυτό θα μίκρινε πολύ η δυνατότητα λάθους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της στην παρατήρηση του ελεκτικού συνεδρίου επιβεβαίωση ότι μια τέτοια δραστική απλούστευση της αποζημίωσης ε, θα, θα μπορούσε πραγματικά να απλουστεύσει τις διαδικασίες και επίσης να δώσει ταυτοχρόνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους ε, δικαιούχους ε, καλύτερη και μεγαλύτερη βεβαιότητα δικαίου και οικονομική βεβαιότητα. Ε, αυτό το σύστημα λοιπόν προτάθηκε από την ε, Επιτροπή προς τον ε, νομοθέτη κατά την προετοιμασία του έκτου προγράμματος πλαισίου που θα αφορούσε το 2002 με το 2006, αλλά η πρόταση αυτή τελικά δεν ενεκρίθη. Και επομένως φοβάμαι ότι χάσαμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία τότε. Α επανέλθουμε όμω τώρα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Στην γνωμοδότηση της πρώτης, ε, ε, πρώτου 2006 επί του 7ου προγράμματος πλαισίου το ελεγκτικό συνέδριο καλωσόρισε τι προτάσει απλούστευση των οικονομικών συστημάτων. Το ελεγκτικό συνέδριο θεώρησε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως θα έπρεπε να αποσαφηνίσει τους ε, κανόνες συμμετοχής, δηλαδή να αναφέρεται σαφώς στους τύπους δραστηριότητας, στους τρόπους ειδικέ ειδικέ δραστηριότητες και τύπο ε, κόστου, αν θα είναι άμεσο ή έμεσος, ε, αν θα είναι κατά αποκοπήν κτλ. Και επανέρχομαι εδώ στου προηγούμενου ομιλητέ, δηλαδή ότι η πρόταση ήταν και δικιά σας και επομένως ε, ε, κάλυπτε και κάποιες ανάγκες του δικού σας οργανισμού. Κατά την άποψη της, ε, του ελεκτικού συνεδρίου, η νομική βάση θα έπρεπε να είναι πιο σαφής και επομένως να δίνει νομική ασφάλεια στους συμμετέχοντες όσον αφορά τους, οικονομικού τους οικονομικούς κανονισμούς ήδη από το 7ο πλαίσιο. Ας πούμε, ε, όσον αφορά του, τους, ε, τις καταποκοπήν ε, αμοιβές. Um, Uh, Όσον αφορά λοιπόν τις καταποκοπήν ε, αμοιβέ, ε, το ελεγκτικό συνέδριο ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν σαφώς καθορισμένες δέσμες εργασίας για κάθε πρόγραμμα και επομένως εδώ δεν υπάρχει διάσταση απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέτοιου είδους καταποκοπήν κόστη θα πρέπει να καθορίζονται και με βάση βεβαίως μια ενδελεχή διαδικασία διαπραγμάτευσης. Και ξέχασα να σας πω ότι το πρακτικό πρόβλημα προκύπτει τη στιγμή που, αθρηστικά, που, γίνονται οι τελευταίες αθροίσεις και επομένως προχωράμε στις ε, τελευταίες ε, πληρωμές και ε, πρέπει να πω ότι εκεί είχαμε πρόβλημα όταν είχαμε ε, δραστηριότητες οι οποίες αφαιρέθηκαν την τελευταία στιγμή, όταν είχαμε τροποποίηση της ε, διαπραγμάτευσης κτλ. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι ναι, από τη δική σας πλευρά λέτε ότι θα πρέπει τα πράγματα να λυθούν, αλλά και από τη δική μας πλευρά βλέπουμε ότι όταν υπάρχουν πολλές αλλαγές και εμείς πρέπει να προσαρμόσουμε τους υπολογισμούς μας. Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα και να ασχοληθούμε με άλλα ζητήματα των δαπανών για λόγους έρευνας αλλά βεβαίω ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχω και τον χρονικό περιορισμό. Ε, να πω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει όλες τις πληροφορίες που έχουν ε, συλλεγεί για την πιστοποίηση των, της μεθοδολογίας τιμολόγησης από την πλευρά των δικαιούχων έτσι ώστε να ε, ε, υπάρξει μια σωστή οριέα ε, βάση για τα προσωπικά κόστη και τα οποία μπορεί να πιστέψει κανείς ότι βασίζονται στο πραγματικό κόστος. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε από τη στιγμή που το προσωπικό κόστος αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού κόστους το οποίο συνήθως αναφέρουν οι δικαιούχοι. Και πρέπει να σας πω ότι και όταν εργαζόμουν στην ε, Γερμανία αντιμετωπίσαμε και τότε τέτοιου είδους προβλήματα και σαν μέλος της, του ελεγκτικού συνεδρίου υπεύθυνο ε, για, την, ε, ε, για την εργασία που αφορά την δήλωση αξιοπιστίας, την DAS, όσον αφορά την πολιτική ενέργεια. Μπορώ να σας πω ότι εδώ και τρία χρόνια έχουμε κάποια προβλήματα τα οποία τα έχουμε υποβάλει σχετικά με το, πρόγραμμα, με το και το 7 πρόγραμμα πλαίσιο. Ε, έχουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία ε, σας υποβάλλουμε. Στην ετήσια αναφορά του 2007 το Συμβούλιο επανεισάγει την σύστασή του για απλούστευση και αποσαφήνιση των κανόνων υπολογισμού και αναφοράς ε, κόστους από τους ε, δικαιούχους ε, και να χρησιμοποιείται το καταποκοπήν ποσό όπου και όσο περισσότερο γίνεται. Στην ετήσια έκθεση του 2008 αναφέρεται ότι στα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσε τα συστήματα ελέγχου και απλούστευσε τους κανόνες ε, ε, χρηματοδότησης ε, των προγραμμάτων έρευνας. Αυτά τα μέτρα συνέβαλαν στην μείωση του επίπεδου λάθους για αυτήν την ομάδα στρατηγικής, έτσι ώστε να διατηρηθούν αυτά τα θετικά αποτελέσματα και η θετική τάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε πρώτον να διασφαλίσει την αυστηρή εφαρμογή των ελέγχων, κυρίως δε αυξάνοντας την αξιοπιστία των πιστοποιήσεων οικονομικών ελέγχου και ε, επίσης δεύτερον ε, ευθυγραμμιζόμενοι με τις ε, πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τους γενικούς δημοσιονομικούς κανόνες να ε, απλουστευθούν ε, περαιτέρω οι κανόνες ε, χρηματοδότησης για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο, το υπαριθμόν 8, διατηρώντας ταυτοχρόνω το στόχο ενός ελέγχου αποτελεσματικού του κόστους και της αποτελεσματικότητας. Όσον αφορά τώρα το μέλλον. και έτσι ώστε να αποφύγουμε περί τους κινδύνους και επιπλέον ε, κόστος λόγω των ελεγχών. Των ελέγχων, συγγνώμη. Πιστεύουμε ότι η έλεγχοι αυτή θα πρέπει να είναι καλύτερα προσαρμοσμένη ε, ε, το επίπεδο, ε, το επίπεδο ανοχής όσον αφορά τον κίνδυνο είναι μια πολιτική απόφαση που πρέπει να συζητηθεί εδώ στο Κοινοβούλιο και πρέπει να συζητηθεί μεταξύ ας πούμε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν ε, αποτέλεσμα της ε, ε, διαπραγμάτευσης, της συζήτησης αυτής ε, είναι ε, το επίπεδο κινδύνου, το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου να ψηλώσει, να μεγαλώσει εμείς σαν ελεκτικό συνέδριο δεν θα έχουμε κανένα λόγο σε αυτό. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα λογικό κατόφλι κινδύνου και εν πάση περιπτώσει εμείς έχουμε έναν σαφή οδικό χάρτη. Για μας υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου του κινδύνου που είναι σαν τους φωτεινούς σηματεδότες ε, του ελέγχου κυκλοφορίας. Δηλαδή ε, το κόκκινο είναι πάνω από 5, το ε, κίτρινο είναι μεταξύ 2 και 5 και το πράσινο είναι κάτω από 2. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Εμείς δεν ερμηνεύουμε με τρόπο διαφορετικό, τον τρόπο, με, τρόπο διαφορετικό συγγνώμη, το πώς μπορούμε να δεχτούμε τις δαπάνες. Επιτρέψτε μου να προσθέσω και κάτι τελευταίο. Κάποιες από τις παρουσιάσεις και κάποια από τα επιχειρήματα τελείωσαν ε, κάνοντας κάποιες προτάσεις δημιουργίας νέων φορέων, νέων οργανισμών κτλ. Νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε κάθε ενδεχόμενο. Αλλά εάν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι στην ουσία εμείς συζητούμε για απλούστευση και για μείωση των ε, υπαρχόντων φορέων στην ουσία. Ε, το να δημιουργήσουμε νέους φορείς για να απλουστεύσουμε παλιές διαδικασίες ε, νομίζω ότι είναι λίγο παράδοξο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χάραλντα Νόακ από το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα έχουμε τώρα δυνατότητα συζήτησης με τους ε, βουλευτές. Δίνω το λόγο στον κύριο Ντί. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μας είπε ο προσκεκλημένος μας που μας βοηθούν να αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε στο μέλλον. Τώρα, λίγο γρήγορα, πώς έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Στην προηγούμενη θητεία της η Επιτροπή μέσω του Πρόεδρου Μπαρόζο ε, ζήτησε μια θετική δήλωση εξοπιστίας που δεν επετεύχθη. Και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θυμόντουσαν βέβαια πολύ καλά την ε, ε, καθαίρεση της Επιτροπής Σαντέρ, αλλά δεν θέλαμε να δώσουμε και τσέκαν λευκό. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί λοιπόν ελέγχου που μέσω διαφορετικών ερμηνιών των εξάντε αναλύσεων της χρηματοδότησης είχαν σαν αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε φτάσει σε μια δύσκολη κατάσταση και δύσκολες σχέσεις ανάμεσα στα σε εκτιμήσει των ευρωπαϊκών οργάνων και το τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο, Κυρίω λόγω των εθνικών μηχανισμών. Πρέπει να ξεφύγουμε από το παρελθόν. Υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί που εμποδίζουν τα πράγματα να προχωρήσουν. Λυπάμαι λοιπόν πολύ που είμαστε στην κατάσταση που είμαστε. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από την Όλαφ που δημιουργούν ένα δύσκολο κλίμα στο όλο θέμα. Θα ήθελα να το συζητήσουμε μεταξύ Ευρωβουλευτών, Πρόεδρε, και θα τελειώσω με αυτό. Πρέπει να ξαναδούμε όλα τα εξαίρετα αυτά στοιχεία τα οποία σήμερα ακούσαμε και πρέπει να βγούμε από αυτήν την νομική αβεβαιότητα που επικρατεί και στην Επιτροπή πέντε χρόνια μετά από την τελευταία πληρωμή να ψάξει να βρει τα λάθη με έναν τρόπο πιο αξιόπιστο. Και επιμένω, και τελειώνω με αυτό, για το ότι πρέπει να βρούμε τα διοικητικά μέσα, τα οικονομικά μέσα, τις κατάλληλες πολιτικές, ώστε να ξεφύγουμε από το παρελθόν. Οι ερευνητικοί οργανισμοί κάνουν ε, ελέγχους πάνω στους ελέγχους. Σίγουρα μπορεί να υπάρξει ανάγκη για διαιτησία. Αλλά πρέπει να ξεφύγουμε από τις καταστάσεις του παρελθόντος και εκφράζω την επιθυμία οι δικαιούχοι που πήραν το λόγο σήμερα το πρωί όλοι ενωμένοι να συμφωνήσουν με την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού στον οποίο θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Grazie. Ευχαριστώ. Άλλες παρεμβάσεις. Η κυρία Τόγια. Πρέπει να πω ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να κινηθεί κανείς στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, έστω και αν ασχολούμαστε ε, με το ίδιο θέμα όλοι, γιατί ε, ε, δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε ποιο πρέπει να κάνει τι. Δηλαδή εδώ συζητάμε, λέμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν, αλλά δεν ξέρουμε ποιο πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα. Η εκπρόσωπο της Ισπανικής ε, Προεδρίας μα είπε ότι στο Συμβούλιο θα προωθηθεί ένα έγγραφο αλλά δεν κατάλαβα γιατί εκεί δεν θα αναφέρεται η πρόταση αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα πρώτο βήμα. Και εγώ θα ζητήσω από τον πρόεδρο της δικής μου επιτροπής εάν μαζί με την Προεδρία μπορεί να κάνει μια μικρή task force έτσι ώστε να βγούμε από αυτή την ε, αγχωτική κατάσταση ε, όπου εμείς μιλάμε αλλά είναι λίγο έπερα απτερόεντα, τα παίρνει ο άνεμος και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα το οποίο πραγματικά θα είναι αποτελεσματικό. Και να πω το εξής. Συμφωνώ με την τελευταία παρατήρηση του τελευταίου παρεμβαίνοντος. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι είναι αρνητικό το να σκεφτούμε τη δημιουργία νέων φορέων που θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την, ε, ε, την ε, πολυπλοκότητα και τη διαφοροποίηση των ερμηνεών. Μα δεν είναι δυνατόν για να απλουστεύσουμε για να να κάνουμε ένα νέο νόμο για την απλούστευση ή να δημιουργήσουμε μια νέα δομή που θα δουλέψει και θα κάνει προτάσεις για την απλούστευση. Ε, και μερικές φορές διαπιστώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι φοβούνται την απλούστευση γιατί φοβούνται ότι θα υπάρξει ένας νέος νόμος που στο όνομα της απλούστευσης θα δημιουργήσει νέους κανόνες που θα, θα διαγράψουν όλους τους παλιούς και επομένως η δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα θα πρέπει να διαγραφεί και να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάλι για το μέλλον. Φοβούνται λοιπόν όταν ε, ε, διαπιστώνουν ότι ή μάλλον όταν φοβούνται ότι θα υπάρξει νέο ε, κανονιστικό πλαίσιο, νέα στοιχεία. Τώρα λυπάμαι βέβαια και εγώ που δεν είναι σήμερα εδώ η Όλαφ μαζί μας και ελπίζω ότι τελικά από όλη αυτή τη συζήτηση θα απορρεύσει κάτι θετικό. Πιστεύω ότι θα υπάρχει η στήριξη του Κοινοβουλίου. Αλλά και το Κοινοβούλιο όπω και τα άλλα θεσμικά όργανα θα πρέπει να αποφασίσουν ότι θα κάνουν ένα βήμα προ αυτή την κατεύθυνση. Εάν και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και το Συμβούλιο κάνουν ένα βήμα τότε πραγματικά θα είμαστε ε, ενεργά υποκείμενα, θα κάνουμε μια ενεργή πρόταση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιάλα Σέντερ. <clears throat> Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω και εγώ να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ακρόαση. Στην ε, Επιτροπή του Ελέγχου Προπολογισμού το θέμα του ανεκτού σφάλματος ήταν κάτι που μας ε, απασχολεί συνέχεια. Τώρα στο έκτο πρόγραμμα, στο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν υποφεληθήκαμε, δεν υποφεληθήκαμε αρχικά αρκετά. Το Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, δεν είχε τις ίδιες δυνατότητες που έχει και σήμερα. Όμως, μπορούσαμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Και αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Να έχουμε πολιτικές συμφωνίες και η Ισπανική Προεδρία το φροντίζει για αυτό το θέμα. Οπότε οι προτάσεις που εξετάζει το Συμβούλιο είναι καλές περιμένουμε και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας βοηθήσει. Αλλά εννοείται, κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, το μπαλάκι είναι στο δικό μας γήπεδο. Εμείς είμαστε ο νομοθέτης, οπότε συμφωνεί σε αυτές οι πολιτικές που πρέπει να γίνουν για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Η ζήτηση που υπάρχει από τον ερευνητικό κόσμο είναι το κεντρικό στοιχείο. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Από την άλλη μεριά και από τους ερευνητές πρέπει να ζητάμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Εγώ προέρχομαι από τον κόσμο των πανεπιστημίων και ξέρω, έχω δουλέψει και συνεργάζομαι με τους ε, συναδέλφους μου από το πανεπιστήμιο. Πρέπει λοιπόν από τα πανεπιστήμια, από την κοινωνία της έρευνας να το ζητήσουμε αυτό περισσότερο. Είναι πολύ βασικό να υπάρχει τέτοια διαφάνεια, όχι τόσο για μας, όσο για τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει μήπω ε, να απαντήσει κάποιος από τους εισηγητές, η κυρία Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω μόνο να διευκρινίσω κάτι για να μην υπάρχει σύγχυση μετά από αυτά που είπε η κυρία Τόγια. Εγώ αναφέρθηκα στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει την πρότασή της για τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού και προβλέπεται αυτό για τα τέλη Μαΐου. Και γι' αυτό ακριβώς η Ισπανική Προεδρία δεν θα μπορέσει να χειριστεί αυτό το ζήτημα. Θα είναι, φαντάζομαι, αντικείμενο της Βελγικής Προεδρίας. Στο Συμβούλιο προς αυτή την γραμμή πάμε. Η ανακοίνωση για την απλοποίηση δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Σήμερα ε, πρόκειτο να εγκριθεί από το Σώμα των Επιτρόπων, στη συνεδρίαση δηλαδή των Επιτρόπων. με διάφορα στοιχεία υπέρ της απλοποίησης του προγράμματος πλαίσιου. Εποφελούμε από αυτή την ευκαιρία για να σας πω και κάτι ακόμα, ότι εδώ και καιρό είμαστε στον ίδιο δρόμο, όπου προστίθενται δυσκολίες αντί να Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθήσουμε, όπως λέει και η κυρία Τόγια, η προσπάθεια απλοποίησης που κάνουμε να μην περιπλέξει τη ζωή των δικαιούχων και των ερευνητών. Είναι πολύ βασικό για μας να λαμβάνουμε υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία όταν σχεδιάζονται καταρχήν τα προγράμματα και σχεδιάζονται και οι σχετικοί διαγωνισμοί για τις αιτήσει. Θέλουμε να διευκολύνουμε τη ζωή του κόσμου και όχι να την δυσκολέψουμε και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί έχοντας υπόψη μας το ότι η Ευρώπη πρέπει να εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νόκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι στόχοι και η σκοποί αυτοί ε, θα συνεχίσουν να επιδιώκονται, ότι θα συνεχιστεί προσπάθεια απλοποίησης. Το ελεγκτικό συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι διατεθειμένο να συμμετάσχει στην διαδικασία αυτή. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μία πτυχή του θέματος που τέθηκε στη συζήτηση. Έγινε μια αναφορά ε, στις ε, παγκόσμιες αρχές, ε, προδιαγραφές, τι λογιστικέ, δηλαδή, γνωρίζετε υπάρχει το ε, οι δύο ε, πλευρές, δηλαδή αμερικανική και γερμανική, που ε, ψάχνουν να βρουν μία, ε, κάνουν μια προσπάθεια τυποποίησης των ε, κανόνων αυτών. Η κυρία Ντελατόρε. Εγώ επιβεβαιώνω ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα εγκριθεί την επόμενη Πέμπτη, γι' αυτό και σήμερα δεν μπόρεσα βέβαια να σας την παρουσιάσω, αλλά υπενθυμίζω σε όλους και όλους μας ένα πράγμα, ότι θα κατατεθούν επιλογές με την ανακοίνωση αυτή, γιατί όχι λύσεις, τουλάχιστον σύμφωνα με την δημόσια διαβούλευσή μας, δεν σημειώνεται ομοφωνία για τις λύσεις. Ορισμένοι προτιμούν ένα σύστημα βασισμένο, όπως ακούσαμε και σήμερα το πρωί, στο πλήρες κόστος και πραγματικό κόστος του συστήματος των project. Άλλοι προτιμούν ε, να επικεντρωθούν μονάχα στα αποτελέσματα, Άλλοι προτιμούν καταπικοπήν ποσά για ολόκληρη την Ευρώπη, άλλοι πάλι προτιμούν, προτιμούν ε, scales of, of unit, ε, οι κλίμακε μονάδων. Υπάρχει λοιπόν μια ποικιλία διαφόρων ε, βημάτων. Η Προεδρία είπε ότι βρισκόμαστε ακόμα στην διαβούλευση. Όλες οι, έχουν, όλες οι λύσεις έχουν κάποια θετικά σημεία. Πάντως εσείς ως νομοθέτης θα πρέπει να κάνετε επιλογές. Επιλογές που καμιά φορά μπορεί να είναι και οδυνηρές, εφόσον πάντως όλοι επιθυμούμε να επιτύχουμε το στόχο της απλοποίησης. Ευχαριστώ πολύ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα δώσω το λόγο στον Άλντο Πατριτσέλο, εισηγητή της Επιτροπής μας. Ήταν εξαιρετική αυτή η σημερινή συζήτηση. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την γραμματεία της Επιτροπής που με όρισε ε, η συγητή Και ήμουν και παλιότερα ε, σαν αντιπρόεδρος της ε, Ήτρε, μέλος της ομάδας που εκπώνησε τις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ όλους ε, για τη σημερινή συζήτηση, ιδιαίτερος δε ευχαριστώ τον Πρόεδρο, ο οποίος ενστερνίστηκε την πρόταση του 2009, όταν δηλαδή είχε αποφασιστεί να οργανωθεί η ακρόαση αυτή για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο με διτό στόχο πρώτον να καταδειχθούν οι ιδιαιτερότητες του προγράμματος και τα σημεία τα οποία προκάλεσαν προβληματισμό των, τα προηγούμενα χρόνια και δεύτερον να προετοιμαστούν τα επόμενα προγράμματα πλαίσιο κάποιες γενικές θεωρήσεις. Η πολιτική ενέργεια της Ευρώπης βρίσκει την βάση της στο 132 των συνθήκων που προβλέπει ότι τα προγράμματα έρευνας θα πρέπει να διασφαλίζουν την τεχνολογική πρόοδο της Ευρώπης. Υπάρχουν, ε, δαπάν, ε, υπάρχουν ε, πιστώσεις πολυετής για την χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής έρευνας. 24 δις ε, θα έχουν στη διάθεσή της ε, τα ερευνητικά κέντρα ε, βάσει του 7ου προγράμματος πλαισίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρόκειται για δημόσιο χρήμα το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ορθά. Σύμφωνα με τη συνθήκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των προγραμμάτων και την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών και των αποτελεσμάτων. Όμως η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται βάσει της στοχοθέτησης. Η παρακολούθηση ε, συνεπάγεται και την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Όσον αφορά την αξιολόγηση, πιστεύω ότι, και αυτό αποδεικνύεται βεβαίως και από την συζήτηση, ότι χρειάζεται μια καλύτερη, σαφέστερα διατυπωμένη ε, στρατηγική αξιολόγηση ε, η οποία θα πρέπει να ε, αποτελεί κοινή βάση των ερευνητικών προγραμμάτων και βεβαίως θα πρέπει η αξιολόγηση να γίνει κατά κάποιο τρόπο μια ενδιάμεση οδός ανάμεσα στα προγράμματα και τους στόχους τους και τα τελικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Όσον αφορά την εποπτεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ορίσει μία περιορισμένη αλλά πάντως σαφή σειρά δικτών αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ξεκινώντας από, το, από τα παλαιότερα προγράμματα πλαίσιο, η παρακολούθηση γίνεται από μια ομάδα εξωτερικών ε, εμπειρογνωμόνων. Αλλά ε, εδώ υπάρχουν προβλήματα. Αυτές οι ομάδες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων συνεδριάζουν ε, όχι πολύ συχνά και πρόκειται για ομάδες οι οποίες συστήνονται ad hoc και συνήθως το αποδεκτό, το, το, το, τελικό επίπεδο χρηματοδότησης είναι χαμηλότερο από αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν, να δημιουργηθεί ενδεχομένως μια ευρωπαϊκή ομάδα και να δοθεί περισσότερη να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στις ad hoc επιτροπές αποτελεσματικότερη διαδικασία όσον αφορά τις τεχνολογίες και τις αξιολογήσεις. Πέρα από τις ευρωπαϊκές αξιολογήσεις γίνονται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δηλαδή, γίνονται και οι αξιολογήσεις σε επίπεδο κρατών μελών. Αυτές ε, οι εθνικές αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνονται βάσει κοινή ορολογίας και κοινή μεθοδολογίας. Έτσι λοιπόν, ε, ε, ώστε να μην δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα εις τους δικαιούχους οι μεθοδολογικές δυσκολίες ε, που αντιμετωπίζουμε για την αξιολόγηση των προγραμμάτων έγκυται σε χρονικά προβλήματα, προβλήματα δηλαδή ε, χρόνου, προβλήματα τα οποία συνδέονται με την ίδια την φύση της ερευνατικής δραστηριότητας, άρα ε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο συγκερασμού ε, των προβλημάτων της έρευνας αφενός, προγραμματισμού της έρευνας αφετέρου και ε, χρονοδιαγραμμάτων οικονομικών κατά τρίτο λόγο. Θα πρέπει να υπογραμμιστούν τα στοιχεία τα οποία αφορούν ερευνητικά προγράμματα που είναι πιθανό να κρατήσουν περισσότερο από το αρχικά προβλεπόμενο. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε ε, και για τους, να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά ε, το, τον οικονομικό, δημοσιονομικό κανονισμό για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ε, δηλαδή, καθυστερήσεις όσον αφορά τις εκτονιστέρων, τους εκτονιστέρων υπολογισμούς και ελέγχους. Επίσης, θα πρέπει να αποσαφινιστούν περαιτέρω και να δημοσιοποιούνται όλοι οι κανονισμοί πριν ξεκινήσει η προκήρυξη. Σύμφωνα με την ε, προκήρυξη και λαμβάνοντας υπόψη την περιπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου ε, θα πρέπει να ε, κατανοήσουμε ότι δημιουργούνται επιπλέον βαριά κόστη η ανάγκη περαιτέρω απλούστευσης στην διαχείριση των προγραμμάτων γενικότερα και των μεμονωμένων προγραμμάτων ειδικότερα. Το κόστος του προσωπικού ε, των ελεγκτικών προγραμμάτων ε, στα ε, που προβλέπεται από την προκήρυξη. Η καθυστερημένη δημοσιοποίηση της προκήρυξης μονάχα περισσότερα προβλήματα δημιουργούν στα ερευνητικά κέντρα. Άλλο σημαντικό πρόβλημα, η διαφορετική ερμηνεία του δημοσιονομικού κανονισμού ε, από τα εμπλεκόμενα μέρη η ανάγκη που κατά την άποψή μου υπάρχει να δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία θα είναι σε θέση ε, με έναν ε, ενιαίο τρόπο ερμηνείας να ερμηνεύει όλες τις ε, διαφορές οι οποίες προκύπτουν. Άλλο σημαντικό θέμα, η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους δικαιούχους όσον αφορά αλλαγή των κανόνων. Τέλος, το, η μείωση του διοικητικού βάρους έτσι ώστε να μπορούν ε, και μικρότερες ερευνητικές μονάδες ε, να συμμετέχουν και επίσης να μην αποθαρρύνονται τα ερευνητικά κέντρα ή τα πανεπιστήμια από το να ε, συμμετέχουν στις, στις διαδικασίες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι κάποια πρώτα στοιχεία τα οποία ε, μας οδηγούν ε, στο ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο πιο ασφαλές, ε, ένα πλαίσιο το οποίο θα, θα γεννήσει την εμπιστοσύνη των εμπλεκομένων, είτε πρόκειται για ερευνητικά κέντρα, είτε πρόκειται για παρεπιστήμια είτε πρόκειται για επιχειρηματίες. Θα τους δώσει λοιπόν την εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά προγράμματα έτσι ώστε να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδικασίες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και επίσης να δώσουμε και τη δυνατότητα πρόσβασης στα προγράμματα αυτά των μικρότερων και λιγότερο δυνατών επιχειρήσεων. Αυτή η απλούστευση λοιπόν είναι απαραίτητη γιατί είχαμε μία εικονική απλούστευση ε, μέχρι τώρα και επομένως ε, χρειαζόμαστε μία πραγματική απλούστευση η οποία δεν θα προκαλεί περαιτέρω προβλήματα στις μικρές ερευνητικέ μονάδες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Άλτο Πατριτσέλα, τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ και την εκπρόσωπο της Επιτροπής, του Συμβουλίου και ε, του ενεκτικού Συνεδρίου που μας ε, μίλησαν για θέματα τα οποία μας είναι ιδιαίτερως προσφυλή. Οτιδήποτε σχετίζεται με τα πανεπιστήμια, με την έρευνα, με την ανάπτυξη ε, μας είναι ιδιαίτερος προσφυλές. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος άλλος να πάρει τον λόγο. Να υπενθυμίσω ότι δεν έχουμε άλλα σημεία στη μερήσα διάταξη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Την Δευτέρα 31 Μαΐου, 3 ε, το μεσημέρι, θα έχουμε την επόμενη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ.